So, good afternoon. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Απασχόλησης. Πρώτο σημείο της μίας διάταξης, έγκριση. Έχουν γίνει οι αιτήσει για τις εξής αλλαγές. Ανακοινώσεις της Προέδρου θα έλαβουν χώρα αμέσως μετά την ψηφοφορία. Έπειτα το σημείο 4 για το σχέδιο ψηφίσματος για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα το εξετάσουμε τελευταίο, λίγο πριν την ψηφοφορία, και το σημείο 12, Οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων, θα το εξετάσουμε μετά το σημείο 6. Το σημείο 21. Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Απασχόλησης στο Λονδίνο θα εξεταστεί μετά το σημείο 12, αν μας επιτρέψει ο χρόνος, και η ψηφοφορία Έπειτα θα αρχίσει στι 4 και 4, θα για τι 4. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει για την ημερήσια διάταξη, μπορεί εκείνη να εγκριθεί, να εγκριθεί με τι τροποποίησει που μόλι σα ανακοίνωσα. Τώρα, στα εγγραφά σας μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά τη συνεδρίαση ε, του Ιουλίου και εκείνη του Σεπτεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά χωρί τροποποίηση. Περνάμε τώρα στο σημείο 5, μέτρα που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Η συνάδελφός μας Edith Bauer είναι η συγγήτρια. Εδώ εξετάζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες που λάβαμε για το σχέδιο έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας. Οι επιτροπές ΛΥΜΠΕΦΕΜ και ΠΕΤΗ αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν. Έχουμε 173 τροπολογίες. Έχουν προταθεί 39 συμβιβαστικέ τροπολογίες από τον κυρία Μπάουερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η οδηγία αυτή που εστιάζει στην καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση την ηθογένεια Είναι μια οδηγία που σκοπεύει να εφαρμόσει τον κανονισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, επειδή υπάρχουν σαφείς περιορισμοί στο, εύρος, ε, στο πεδίο εφαρμογής της ε, οδηγίας και θα ήθελα να αναφέρω κάποια ζητήματα τα οποία έχουν συζητηθεί πολύ συχνά. Τρία από αυτά όσον αφορά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Η οδηγία αυτή μετά από τον κανονισμό αποκλείει τις αλληλοεπικαλύψεις με τον κανονισμό 883 για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η οδηγία αφορά μόνο τα κοινωνικά πλεονεκτήματα μια διαφορετική κατηγορία από εκείνη της κοινωνικής ασφάλισης. Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τώρα, που είναι και το δεύτερο σημείο που συζητήθηκε, ε, η κατάσταση έως τώρα έχει ως εξής. Πολύ συχνά, σε περιπτώσεις διασυνοριακών εργαζομένων, οι διακρίσεις ε, με βάση την ηθαγένεια αποφεύγονται και αντί αυτές ε, σημειώνονται διακρίσεις ε, με βάση τον τόπο κατοικίας. Το Συμβούλιο οδεύει και εκείνο προς ε, την ίδια κατεύθυνση και πολλές φορές ε, συναντάται μία κάπως ε, περίεργη διατύπωση η οποία προκύπτει από τα διαφορετικά νομικά συστήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Σε ορισμένα από αυτά ορισμένα βασίζονται στις αποζημιώσεις Άλλες όμως χώρες όπως η Δανία έχουν περιπτώσεις όπου τα συνδικάτα μπορούν να αναλάβουν δράση εκπροσωπώντας τα συλλογικά συμφέροντα αυτεπάγγελτα. Ορισμένες ε, φορές λοιπόν χρησιμοποιούμε τη διατύπωση as appropriate και θα ήθελα να εξηγήσω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούμε μια τέτοια διατύπωση ή όπως ισχύει στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Καταρχάς, ε, μαζί με τους εσκιώδεις εισηγητές να πω ότι προσπαθήσαμε πολύ να έρθουμε σε έναν συμβιβασμό για το θέμα αυτό. Και θα ήθελα επίσης, εκτός από τους εσκιώδεις συζητητές, να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την ε, πολύτιμη, χρήσιμη και αποτελεσματική βοήθεια που παρήχαν. Και να ευχαριστήσω επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εκπρόσωποι της οποίας ήταν στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε διευκρίνηση όσες φορές ε, την ε, ζητήσαμε, όσες φορές συναντήσαμε προβλήματα και χρειαζόμασταν επιπλέον διευκρινήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κρίστιανσεν. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Μπάουερ. για την εξαιρετική συνεργασία. Έπρεπε να κάνουμε πολλή δουλειά σε πολύ λίγο χρόνο και ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αυτή η καλή συνεργασία την οποία και είχαμε. Θα ήθελα να, το, να αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία τα θεωρώ επιτεύγματα. Καταρχάς είναι πολύ σημαντικό ότι η οδηγία αυτή είναι μια οδηγία για τους εργαζόμενους και θα εξασφαλίσει τα δικαιώματά τους, την κινητικότητά τους και την ίση μεταχείρισή τους. Οπουδήποτε και αν επιλέξουν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κοιτάξουμε τώρα τις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες, στις ε, προκλήσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές φορές οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα σύνορα, θα δούμε ότι η οδηγία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τους υφιστάμενους κανόνες για ελεύθερη μετακίνηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νέες δομές να μην παρακολύσουν το έργο των ε, υφιστάμενων οργανισμών, διότι η δημιουργία περισσότερων οργανισμών θα δημιουργήσει περισσότερη σύγχυση. Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις που θα παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς απολαβές. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης οι εργαζόμενοι να έχουν δελτία μισθοδοσίας ε, απολύτως κατανοητά. Υπάρχουν τώρα κάποιοι άλλοι συμβασμοί που δεν μπορώ να τους ε, δεχτώ. Ένας από αυτούς που έρχεται από την ίδια την κυρία Μπάουερ και στηρίζεται και από το ΕΛΚ. Ο συμβιβασμός αυτός αφορά το σημείο 29 στον συμβιβασμό 8D. Αναφέρεται ένα παράλληλο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης και αυτό είναι κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει νομική δυνατότητα για κάτι τέτοιο αλλά πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα άλλο καθεστώς ε, πέραν των 28 υφιστάμενων καθεστώτων στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να παρατηρήσω ότι βλέπω κάποιες ομοσπονδιακές ε, τάσεις και το θεωρώ κάπως προβληματικό. Θα ήθελα λοιπόν να συστήσω να καταψηφίσουμε την συμβαστική αυτή πρόταση. Ωστόσο να πω ότι υπήρξε εξαιρετική συνεργασία στο σύνολο της έκθεσης και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ο Φίλιπ Τεπάρκ. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι συντομότατος. Ευχαριστώ την συγκητή. Πολύ καλή συνεργασία. Κινηθήκαμε τάχιστα. Πετύχαμε καλούς συμπιβασμούς. Είναι σαφές ότι αντιμετωπίσαμε πολύ σημαντικό θέμα. Πολλές εταιρείες, μικρές, μεγάλες, αποκτούν όλο και πιο διεθνή χαρακτήρα και επεκτείνονται και στην Ευρώπη. Άρα, σημαντικό είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων και αυτά να ακολουθούν αυτές τις τάσεις. Να έχουν εγγυημένα τα δικαιώματά τους. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι καλά, έχουμε ισορροπημένη έκθεση. Υποστηρίζουμε τα διάφορα σημεία στη ψηφοφορία, εκτός από τη σημαστική ΚΑΠΑ Λατινικό, που είναι πολύ δύσκολο να τη δεχτούμε. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα όμως, ούτε οι μόνοι βουλευτές που έχουμε πρόβλημα με τη συμβαστική ΚΑΠΑ Λατινικό. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ευρεία συμφωνία στην ψηφοφορία. Είναι σημαντικό να στείλουμε σαφές μήνυμα σαν κοινοβούλιο προς τις επιχειρήσεις και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων και ελπίζω αργότερα στην ψηφοφορία να πετύχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Η Αναλίζα. Ευχαριστώ. Κυρία Κορνέλησεν, ευχαριστώ όλους τους και ηγητές. Αυτή η οδηγία δεν αποκαθιστά κάποια από τα θεμελιώδη προβλήματα που υφίστανται με την κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να προστατεύει κάποιους καλύτερα από άλλους. Ελπίζω να είναι πολύ χρήσιμη η προσπάθεια, θα είναι καλύτερα ενήμεροι, θα έχουν κάπου να στραφούν αν είναι θύματα διάκρισης όπως για ένα φορέα, σε έναν φορέα ισότητας, σε συνδικάτο ή κάποιος φορέας μπορεί να προστατεύσει συλλογικά δικαιώματα ομάδων εργαζομένων και στο πιο καινούριο αυτό κομμάτι καταφέραμε να βελτιώσουμε το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη. Ελπίζω ότι στην πράξη θα καλυφθούν όλοι. Έτσι όλοι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανεξάρτητα του τομέα που εργάζονται θα έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Καθώς πρέπει. Κλείνω ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας βοήθησε πάρα πολύ εξήγησε την περιπλοκότητα την νομική κατάσταση που στρέφεται γύρω από αυτή την οδηγία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μουό έχει το λόγο. Είναι εδώ. Ε, merci, Madame la Présidente. Νομίζω ότι δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε. Σίγουρα Πρόκειται περί προτάσεως οδηγίας σημαντικοτάτης, διότι διευκολύνει ε, τους και τα μέλη της οικογένειας που ακολουθούν τους μετακινούμενους από τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι λοιπόν για την υποστήριξη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την προσπάθεια. Και ειδικά ευχαριστούμε και αυτή την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. να δίνουμε το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Να ευχαριστήσω ξανά όλους τους ε, συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Ευχαριστώ τους σκιώδεις που εργάστηκαν σκληρά για την επίτευξη συμβιβαστικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συμβούλους μας. Πράγματι εργάστηκαν πολύ σκληρά και μας βοήθησαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε σήμερα αυτή την έκθεση. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η κυρία Χάρκιν είναι η συγγήτρια. Να σας ενημερώσω για κάτι για τα αποτελέσματα. Ανεπίσημος τριμερής διάλογος έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου, προσωρινή συμφωνία επετεύχθη και ανεκρίθη το πακέτο στις 11 Οκτωβρίου και επί το οποίο απασχόληση θα ψηφίσει σήμερα. Λοιπόν, βασικά σημεία της συμφωνίας, το Ταμείο θα ενεργοποιείται σε περίπτωση απολύσεων που οφείλονται σε παγκοσμιοποίηση ή λόγω οικονομικής και χρηματοστατικής κρίσης ε, δεν θα συμπεριληφθούν ειδικέ διατάξεις για τους αγρότες. Όλες οι συμβάσεις θα καλύπτονται και επίσης ε, σταθερής ε, στις συγκεκριμένες διάρκειας, προσωρινής διάρκειας. 35% του κόστου του πακέτου θα είναι η αμοιβή Προβλέπετε χρονοδιάγραμμα. Η Δημοσιονομική Αρχή θα έχει ένα μήνα και όχι έξι εβδομάδε, χρόνο για να λάβει απόφαση για την κινητοποίηση, για την ενεργοποίηση του Ταμείου αυτού σε κάθε περίσταση. Δεν είναι διαθέσιμη η συγγήτρια. Μου ζήτησε να διαβάσω. Um, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ζητώ συγγνώμη τους συναδέλφους που απουσιάζω τη Επιτροπής, αλλά πρέπει στρέψω στην πατρίδα μου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που καταβάλουν προσπάθειες για τη συνέχιση του Ταμείου. Τρίτον, ευχαριστώ τους Κιώδης και την πρόοδο της Επιτροπής για τη στήριξή τους και την αποφασιστικότητά τους κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων. Πετύχαμε κάποια πράγματα και στο τέλος νομίζω ότι οι διαπραγματευτήσεις αλλαγές βελτίωσαν το χρονοδιάγραμμα, την αποτελεσματικότητα και έδωσαν ευρωπαϊκή υποστεθέμενη αξία στο Ταμείο. Η σημαντικότερη αλλαγή στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η συμπερίληψη ισότιμη γνώση αναγκών για κατάρτιση, παιδεία για εκείνους που είναι κάτω των 30 τις περιοχές ΝΑΤΣ 2 όπου εκεί μπορούν να υπάρχουν απολύσεις και μπορεί να υπάρχουν πρωτοβουλίες για απασχόληση. Το Συμβούλιο ήθελε οι ανάγκε των γειτονικών περιοχών των ΑΤΣΔΙΟ 2, που ήταν επιλέξιμε για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, να συμπεριλαμβάνονται και αυτέ, αλλά διαπραγματευτήκαμε συμβαστική λύση όσον αφορά το θέμα, ούτω ώστε το γεωγραφικό πεδίο να παραμείνει ακέραιο. Με άλλα λόγια, οι επιλέξιμε ανάγκε συνδέονται γεωγραφικά με του απολυμμένου εργαζόμενου. Άλλε αλλαγέ συμπεριλαμβάνουν ενιαίο ποσοστό συγχρηματοδότηση 60%, 10% παραπάνω από το 50% που αρχικά προτάθηκε πολεμήσαμε σκληρά για να προσπαθήσουμε να έχουμε τουλάχιστον διπλό, διπλή ποσοστό σήμεση χρηματοδότηση με χώρες προγραμμάτων ή χώρες που συμμετέχουν στα μη συνοχή. Συμφωνήσαμε όμως με ταινία ενιαίο ποσοστό 60% σε αντάλλαγμα για τη δική μας κόκκινη γραμμή να τίθεται ανώτατο όριο όσον αφορά τις διάφορες επιδοτήσεις 35%. Ήταν κόκκινη γραμμή για μα, διότι ανησυχούσαμε για την προστιθέμενη αξία την ευρωπαϊκή και ανταποκριθήκαμε στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Διαπραγματευτήκαμε μείωση 15% στο επίπεδο των ειδικών επιδομάτων εισμένου χρόνου κάτω από το 50% που πρότειναν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Συμπεριλάβαμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για υποβολή και αξιολόγηση προγραμμάτων αντί ανοιχτής διαδικασίας που ε, ήθελε το Συμβούλιο. Εξασφαλίσαμε ότι όλα τα είδη των συμβάσεων και σταθερά και ορισμένου χρόνου, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, καλύπτονται και την αυταπασχόληση, ακόμα και επιχειρήσεις με ένα άτομο καλύπτονται. Ήρθε το Συμβούλιο να καλύπτουμε εταιρείε με έναν ως δέκα εργαζομένους. Θέλαμε ακόμα και οι ατομικές επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνονται. Δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τους γεωργούς και επέκταση του Ταμείου να καλύπτει απώλειες που δημιουργούνται από οικονομική και χρηματοπιστωτική. Εξασφαλίζεται μάλλον η κάλυψη και αυτών που απολύονται λόγω οικονομικής χρηματοστικής κρίσεως. Θέλει κάποιος συνάδελφος να παρέμβει. Ορίστε. Η κυρία Μπάουερ και μετά η κυρία Κορνέλισον. Κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Χάρκιν και την κυρία Μπερέζ. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ήταν από τις πιο δύσκολες στις οποίες συμμετείχα. Πολύ συχνά είχαμε φτάσει στα όρια. Ετέθη να αμφιβόλο ακόμα και η ύπαρξη του Ταμείου. Η ανεργία των νέων. Θέλαμε κάποια λύση γι' αυτό. Ποτέ δεν συζητήσαμε το θέμα αυτό στα πλαίσια της οδηγίας, αλλά ετέθη ως προϋπόθεση, ως όρος από πλευράς του Συμβουλίου. Να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της αναστέλωσης μειοψηφίας. Ήταν δυσκολότατες οι διαπραγματεύσεις. Δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Βελτιώσαμε τη μορφή του Ταμείου, αλλά συμβιβασμός είναι συμβιβασμός. Καμιά φορά ήταν εξαιρετικά δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και συμβιβασμοί με το Συμβούλιο. Ε, πρέπει να επαναλάβω ότι όλοι που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καταλήξουμε σε κάποιους συμβιβασμούς. Για να πετύχουμε τους καλύτερους δυνατούς συμβιβασμούς. Ήταν πολύ σκληρή δουλειά. Αυτό ήθελα να σας πω. Έπρεπε να σας το πω αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Simplement deux mots euh, Και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι αυτή την ε, σκληρή εργασία, τι προσπάθειε που έχουν γίνει από την κυρία Χάρκιν, διότι δεν ε, ήταν κάτι το δεδομένο ε, τη στιγμή που το σημείο εκκίνησης ήταν η ενδεχόμενη απόρριψη αυτού του πλαισίου όπως ακριβώς ανέφερε και η κυρία Χάρκιν γι' αυτό, ε, δέχομαι αυτά που ελέγχθησαν και τα συμπεράσματα επίσης. Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ε, απόλυτα με τους προλαλήσαντες, ιδιαίτερα με τον κύριο Νταρντέν, διότι ήταν πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση και είδαμε ε, ότι ε, βάλαμε στην άκρη τους αγρότες, αλλά την, το πλαίσιο για τους νέους το δεχτήκαμε και το εντάξαμε και ελπίζω ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν ε, συνετά από όλα τα κράτη-μέλη. Έχει βελτιωθεί το όλο σε σχέση με την τρέχουσα χρηματοδότηση. Ελπίζω να ε, χρησιμοποιηθούν πολύ ε, σωστά και να υπάρχει και καλύτερη στοχοθέτηση προς τους εργαζόμενους που πραγματικά χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Uh, thank you so much. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Η κυρία Χάρκιν σας ευχαριστεί ιδιαίτερα για τη συνεργασία. Ας δούμε το 12 στην ε, ημερήσια διάταξη. σε σχέση με την οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα αποτελέσματα των ε, επιχειρήσεων. Φιλ Μπένιον είναι ο εισηγητής. Και εδώ υπάρχουν 98 τροπολογίες, άρα ε, έχει το λόγο Φιλ. Νομίζω ότι θα το παρουσίασα μετά από την ψηφοφορία, αλλά εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για τις τροπολογίες που συνέταξαν. Ε, υπάρχει σωρία τροπολογιών, οι περισσότερες είναι θετικές, όχι όλες. Τις εξέτασα και θεωρώ ότι περισσότερες ακολουθούν την γραμμή που προβάλλω ε, σε σχέση και με τις συζητήσεις κατά τη σύνταξη της έκθεσης. Επίσης έχω υποβάλει τροπολογίες για να διασαφίσω σημεία τα οποία εφήγησαν μετά από το σχέδιο και μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ και μία δεύτερη παράγραφο μιλώντας για το μέγεθος και το στάτος των επιχειρήσεων που θα ε, επηρεάσει το πρότυπο που θα χρησιμοποιήσουν. Επίσης έχω υποβάλει δύο τροπολογίες για τις ευέλθιστες πρακτικές. Υπ' αυτή την έννοια και με τις τροπολογίες μου, καθώς και τις τροπολογίες των συναδέλφων, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε καλούς συμβιβασμούς ε, για τους ε, περισσότερους τομείς. Ίσως υπάρχουν ορισμένοι δύσβατοι τομείς, αλλά νομίζω ότι θα επέλθει συμβιβασμός ως προς το καθεστώς το 29 που είναι και το πιο διφορούμενο, θα ήθελα να πω ότι ζητάμε μία μελέτη, την εκπόνηση μελέτης από την Επιτροπή για να δούμε κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, καθώς και μία μελέτη αντικτύπου. Δεν ζητάμε να ε, εφαρμοστεί τώρα, θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να δούμε την ε, πρακτική πλευρά του ζητήματος. Δηλαδή αυτό καλύπτει η μελέτη. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι το αρχικό κείμενο έχει διασαφινιστεί και σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς ε, και το καθεστώς σήμανσης δεν θα αλλάξει από αυτό το καθεστώς και πιστεύω ότι έμπρακτα θα έχουμε παραδείγματα για την κάθε ε, επιχείρηση διότι μας ενδιαφέρει καλύτερη ε, διαφάνεια και προσβασιμότητα στις ε, επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ε, διασυνοριακές δραστηριότητες και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε συμβιβασμό. Επίσης, ε, θεώρησαν οι πολλοί ότι αυτό το καθεστώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα Νομίζω όμως ότι υπάρχουν ρήτρες διασφάλισης, δεχόμαστε ότι υπάρχει κίνδυνος, αλλά στην αρχική έκθεση τόνισα ότι θα πρέπει να ορίσουμε όλους τους κινδύνους πριν γίνουν οι οποιασδήποτε δεσμεύσεις. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έρονται οι κίνδυνοι, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε τον κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση. Πιστεύω όμως ότι η έκθεση είναι θετική και συμβαδίζει με τα με τα ε, ευεργετήματα που λαμβάνουμε και βοηθά και την εργοδοσία και τους εργαζόμενους. Η Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρξει σωρία τροπολογιών. Εγώ έχω υποβάλει 35 και θα ήθελα να πω ότι ε, δέχομαι την ε, πρόταση όπως έχει διατυπωθεί, αλλά υπάρχουν και κόκκινες γραμμές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, καταρχήν το πρώτο θέμα αφορά την ε, συμμετοχή των εργαζομένων. Μιλάμε και για χρηματική συμμετοχή, οικονομική συμμετοχή. Πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ε, φωνή, δηλαδή να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης. Και αυτό αφορά και την διαχείριση της επιχείρησης. Θα πρέπει λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και αυτό αφορά και τα συνδικάτα. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή αφορά τους κινδύνους, τους κινδύνους δηλαδή την οικονομική, η χρηματοοικονομική συμμετοχή των εργαζομένων. Ο κύριος Μπένιον μίλησε για τις ευκαιρίες που ε, διαμορφώνονται θα πρέπει όμως να προτείνουμε και οικονομικά ε, δημιουργικά μοντέλα. Εδώ ελοχεύει κάποιος κίνδυνος, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι ε, διατρέχουν κινδύνους. Υπάρχει όμως διπλός κίνδυνος, διότι μπορεί να χάσουν και το κεφάλαιό τους οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ε, δράσουμε με ακρίβεια, διότι η θεματική είναι πολύ καλή, αλλά θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ένα άλλο ε, δύσβατο ζήτημα που έθιξε ο κύριος Μπένιον αφορά το νέο καθεστώς. Εγώ αρχικά είχα πει ότι θα πρέπει να δούμε το όλο ζήτημα πώς ε, διαμορφώνεται, αλλά είπαμε ότι τα διάφορα εθνικά συστήματα απαιτούν την αντιμετώπιση των, των επιφυλάξεων και μια γενικότερη σύνεση. Πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι θα πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις από το 21ο σύστημα. Εγώ αρχικά πίστευα ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει αυτή η επιλογή. Τώρα όμως ε, νομίζω θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος το 21 ο σύστημα. Βεβαίως μπορούμε να ζητήσουμε μία μελέτη σκοπιμότητας από την Επιτροπή για να ρίξουμε φως στα πιο δύσβατα σημεία, αλλά νομίζω ότι δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή για να εισαγάγουμε το 21 ο σύστημα. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι θετικές εμπειρίες, πώς έχουν διαμορφωθεί, έτσι ώστε να υπάρξει η σωστότερη δυνατή, η καλύτερη δυνατή χρήση του συστήματος. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος θα λάβει το λόγο από τους δύο, ο ένας ή ο άλλος. Κανένας. Η Επιτροπή δεν έχει να σχολιάσει το θέμα αυτό. Bien, Σας ευχαριστώ. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού. Α, με συγχωρείτε, ο Φιλ Μπένιον. Ο εισηγητής θέλει να επανέλθει. Ε, εντάχει, να ευχαριστήσω τον κύριο Ρέγνερ για τα σχόλια της. Ήταν η βασική μου συνομιλήτρια για το θέμα αυτό και τα σχόλιά της αντικατοπτρίζουν τα δικά μου. Θα το συζητήσουμε και ελπίζω να φτάσουμε σε καλούς συμβασμούς. Όλα αυτά μου φαίνονται εξαιρετικά και ιδιαίτερα σκόπιμα. Άρα στις 25 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού, 5 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, 6 ε, της ε, πρότασης, πρόταση της πρότασης ψηφίσματος που θα θέλαμε να εγκριθεί το Νοέμβριο σε σχέση με την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Μετά την προφορική ερώτηση που θα υποβληθεί στην Επιτροπή. Θα ήθελα να πω ότι δεν ήμουν παρούσα κατά την προφορική. Λυπάμαι διότι η Επιτροπή δεν συμφώνησε για την προφορική αυτή επί της προφορικής στο Συμβούλιο επειδή πρόκειται για μία ανακοίνωση της Επιτροπής για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ μετά από τρία Ευρωπαϊκά Συμβούλια, όπου εφήγει το ζήτημα. Το θέμα λοιπόν τώρα αφορά την ατζέντα του Συμβουλίου. Ε, λυπάμαι που ε, έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα διότι το βασικό μήνυμα ε, αφορούσε το Συμβούλιο. Όμως με βάση την πρόταση ψηφίσματος η οποία βρίσκεται επιτάπητος, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν υποβληθεί 124 τροπολογίες και χτες με τους υπεύθυνους των ομάδων συντάξαμε 20 τροπολογίες συμβιβασμού που θα μας επιτρέψουν να λάβουμε θέση επί του θέματος αυτού. Όταν δω το πνεύμα που διέπει τις τροπολογίες συμβιβασμού, βλέπω ότι λαμβάνεται υπόψη η θέση της Επιτροπής και επίσης θα επιτελεστεί πρόοδος ιδιαίτερα σε σχέση με τη χρήση των δικτών και η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτούς τους δείκτες, διότι έχει σημασία να υπάρχουν οι δείκτες μόνο όταν χρησιμοποιούνται. Να δούμε τη φτώχεια σε επίπεδο παιδιών ή ανηλίκων και την προσβασιμότητα στην υγεία. Αυτοί είναι δείκτες που μας απασχολούν ιδιαίτερα και επετεύχθη η συμφωνία. Επίσης έχει σημασία να ε, συνεισφέρουμε και στην κατάρτιση αυτών των δικτών. Και εδώ η δράση του Κοινοβουλίου είναι κέρια σημασίας. Δεν θα ήθελα να μπω στις λεπτομέρειες των 20 συμβασμών, θα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρο αυτό. Ευχαριστώ όμως τους υπευθύνου και ελπίζω να υποστηρίξουμε τη Γενική Συμφωνία, διότι πέρα από αυτούς τους συμβιβασμούς, ορισμένες παράγραφοι που υπήρχαν στο αρχικό κείμενο της πρότασης, αποσύρθηκαν ιδιαίτερα η αιτιολογική σκέψη Q. Και οι παράγραφοι 10, 9 και 10. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι τροπολογίες που σχετίζονταν με αυτές τις ε, παραγράφους ε, καταπίπτουν. Η κυρία Κορνέλισεν ε, ζήτησε το λόγο. Αλεχάντρο Θέρκας και οι άλλοι στη συνέχεια. Thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήταν σαφές με το φάκελο αυτό ότι οι απόψεις διαφέρουν πάρα πολύ και ανάμεσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες αλλά και ανάμεσα στις, στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. Τα αποτελέσματα δυστυχώς ε, είναι πολύ πιο αποδυναμωμένα από ό,τι περιμέναμε, από ό,τι ήταν αρχικά και αυτό που θεωρώ περίεργο είναι ότι είχαμε διαφορετικές ε, εκθέσεις αυτό το εξάμεινο και ζητούμε εδώ και δύο χρόνια αυτούς τους δείκτες και τώρα που ε, έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αυτούς τους δείκτες παρατηρείται μία πιστοχώρηση Εντάξει, έχουμε συγκεντρώσει κάποια στατιστικά στοιχεία για την φτώχεια, για την ανεργία και για την ε, αύξηση των ανισοτήτων, όμως ε, χωρίς ε, πράξεις τα στατιστικά στοιχεία δεν χρησιμεύουν. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω πώς, μπορείτε, πώς θα μπορέσουμε να επερασπιστούμε αυτούς τους πολίτες που κινδυνεύουν από φτώχεια. Ωστόσο πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί, διότι πραγματικά διαφορετικά θα ήταν γελίο αν και Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πρωτοπόροι και το Κοινοβούλιο υστερήσει. Δεν είμαι εκπλήσωμε για την απόκληση απόψεων. Αυτή η απόκληση απόψεων είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχει μια συμφωνία. Υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να δοθεί κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Νομισματική Ένωση και υπάρχει και συμφωνία που δεν επιβάλλει επαρκή υποχρέωση στα κράτη-μέλη. Διότι είναι θέμα εθνικών αρμοδιοτήτων σε κάποιου τομεί. Αυτά τα δύο ζητήματα λοιπόν τίθενται. Δύο αντιφάσεις για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Και αυτό είναι και το συμπέρασμα του Συμβουλίου. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν και άλλες συζητήσει πάνω σε αυτό. Καταφέραμε να πετύχουμε κάποιου συμβιβασμού. Οι περισσότεροι συμβιβασμοί μπορεί να στηριχθούν από την ομάδα μα το Ε, το F και το L τα λατινικά δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε, το EF και το L και υπάρχει και ένα σημείο που θεωρούμε σημαντικότατο και θα εξαρτηθεί τελική μας ψήφος από αυτό, αφορά την τροπολογία 109. Για την 109 θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι μου αυτό που προτείνεται και δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε σε αυτό το τομέα ένα ευρωπαϊκό καθεστώς, τουλάχιστον για την ώρα, ένα, ένα επίδομα ανεργίας ευρωπαϊκό. Η 109 λοιπόν, η τροπολογία δεν μπορεί να στηριχθεί που δεν είναι από την ομάδα μας. Ευχαριστώ. Ο Αλεχάνδρος Σέρκας και μετά Φιλίπ Τεμπάκερ. <clears throat> Ευχαριστώ. Ο Αλεχάνδρο Θέρκας, ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να πω. Ε, να πω πριν ε, μιλήσω για την ίδια την πρόταση ψηφίσματος για ένα ζήτημα το οποίο είναι ε, εκρεμές. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε προχωρήσει για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα με το Συμβούλιο, διότι είναι γελίο να μην μπορούμε να έχουμε μία αίσια έκβαση με το Συμβούλιο, τη στιγμή που αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να επιληθούν θα πρέπει λοιπόν έγκαιρα να το δούμε το Νοέμβριο. Αν δεν τα καταφέρουμε το Νοέμβριο, θα πρέπει να ζητήσουμε την παρουσία του Συμβουλίου στη συζήτηση. Και αυτή είναι η οδός που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ως προς την πρόταση ψηφίσματος, χτες βρέθηκα στη συνάντηση για τους συμβιβασμούς Πρόκειται για ένα ε, δύσκολο ε, ε, ζήτημα. Μπορούμε να μιλήσουμε για ποτήρι που είναι κατά το ίμιση γεμάτο ή κατά το ίμιση άδειο, ανάλογα με την προσέγγιση. Πολλές φορές χρειάζεται και να ε, καταπέσουν ορισμένες ε, τροπολογίες, διότι οπωσδήποτε είμαστε επικριτικοί ε, ως προς την έλλειψη ισορροπίας των κοινωνικών και των οικονομικών συνιστώσεων. Το ΕΛΚ δεν δέχεται να προχωρήσει περισσότερο. Γι' αυτό ας πούμε ότι το ποτήρι είναι κατά το ίμιση γεμάτο. Έχει γίνει ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός από την Κομισιόν και μας ενδιαφέρει να βελτιωθεί και το πλαίσιο των δικτών. Το ψήφισμα είναι θετικό, κάναμε μεγάλες θυσίες και δεν φτάσαμε στο τέλος της πορείας μας. Θα δούμε πώς θα είναι και η στάση, πώς θα εξελιχθεί η στάση του ΕΛΚ Εν πάση περιπτώσει, ε, μιλούμε και, μιλήσαμε και για τους αυτόματους σταθεροποιητές και γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε με πλειοψηφία. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι έτσι ώστε να εντάξουμε στην ατζέντα μας αυτούς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εργασία. Ο Φίλιπ Τεμπάκερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για μια καλή και ταχεία συνεργασία. Αυτό αποδείχθηκε και χθε το βράδυ όταν το τι συμβαστικέ απολογίε για το θέμα αυτό. Έχουμε καταλήξει σε ένα σχέδιο ψηφίσματο που το βρίσκω αρκετά εξισορροπημένο. Σίγουρα κάποιοι περίμεναν περισσότερα από αυτό, σίγουρα κάποιοι θεωρούν ότι είναι υπερβολικά ακραίο, όμως εγώ το βρίσκω ισορροπημένο. Χθε κατά τη διάρκεια της συνάντησης των σχεδόν εισηγητών καταλήξαμε στο ότι εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τους περισσότερους συμβιβασμούς. Ο C, ο e ο F, I, ο B και ο U, αυτοί οι συμβιβασμοί είναι ε, συμβιβασμοί που μας βρίσκουν ε, αντίθετους. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, οι τροπολογίε 109 και 124 είναι για την ομάδα μας κόκκινη γραμμή. Πιστεύουμε ότι σε αυτήν την περίοδο οικονομικής κρίσης αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς κινούνται αυτοί οι κοινωνικοί δείκτες, τα κράτη-μέλη, στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, εάν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα. Και είναι επίσης ε, ύψης της σημασίας να καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Σε γενικέ γραμμέ όμω, όπω σα είπα, στηρίζουμε την πρόταση ψηφίσματο. Πιστεύω πω το Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχουμε ένα αίσιο τέλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι για τι ε, συνεισφορές σα που απηχούν τι πραγματοποιηθεί σα διαπραγματεύσει που είναι αβαχόρθε το βράδυ. Θα ήθελα απλώ να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να επανέλθω επί του πλέον επιμάχου σημείου. Υπήρξαν πολλά προφανώς. Το πρώτο ήταν τι θα γίνει συγκεκριμένα όσον αφορά τους δείκτες. Νομίζω ότι το μονοπάτι το οποίο ακολουθούμε δεν είναι εύκολο, είναι δύσβατο, αλλά υπάρχει διάθεση συζητήσεων. Άλλο σημείο όμως υπάρχει όπου κόλλησαν οι συζητήσεις είναι μια αλλαγή προσέγγισης που παρατήρησα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αφορά το θέμα που καλύπτει η τροπολογία 108 των φιλελευθέρων, η κόκκινη γραμμή των διαπραγματεύσεων. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω κάποια πράγματα για την υπόθεση. Νομίζω λοιπόν ότι μέχρι το καλοκαίρι προχωρήσαμε καλά. Προφανώς άλλαξαν τα πράγματα σε κάποιες πρωτεύουσες και οδήγησαν σε αλλαγή θέσεων και εδώ. Αυτή, αυτό το θέμα της ελάχιστη, του ελάχιστου επιδόματος ανεργίας ήταν ένα θέμα που ε, ετέθη για λόγους που έχουν εντοπιστεί, σαφώς. Στην Ευρωζώνη, καταρχάς, λείπουν μηχανισμοί αλληλεγγύης. Γνωρίζω ότι μεγάλες προσπάθειες έγιναν όσον αφορά την αλληλεγγύη τι ούτω τρόπος δόθηκε υποστήριξη στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ισπανία, την Πορτογαλία και όλη η Ευρωζώνη παρέμεινε ακεραίη. Όμως το τίμημα της προσπάθειας αλληλεγγύης δεν πρέπει να υποτιμάται. Γι' αυτό χαιρόμεθα που η Οικονομική και Μεσματική Επιτροπή ξεκίνησε μια διαδικασία αναλύσεως των αποτελεσμάτων των εργασιών της Τρόικα σε κάποιες από τις ε, αναφερθήσεις χώρες. Πέραν από αυτό, τα κενά στη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, δεν καλύφθηκαν από τους μηχανισμούς που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Παραμένουν μηχανισμοί αλληλεγγύης μεταξύ τραπεζών, αλλά όχι αλληλεγγύης όσον αφορά τις επενδύσεις σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με το 6-pack και το 2-pack και το Fiscal Compact ε, εφαρμόστηκαν και διάφορες διαδικασίες ε, κυρώσεων. Λοιπόν, εάν είναι να επιβιώσει η Ευρωζώνη και είναι προς συμφέρον όλης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των 28 χωρών συμφέρον να επιβιώσει, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αλληλεγγύης που θα θεσπιστούν. Ξεκίνησε η συζήτηση. Όσον αφορά την αμοιβαία αντιμετώπιση του χρέους, το μοίρασμα του χρέους πρέπει να συνεχιστεί τροφοδοτήθηκε η συζήτηση από μια ανάλυση που έλαβε χώρα και το ακούσαμε στην ακρόασή μας για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού. Ακούσαμε την ανάλυση που αντλεί μαθήματα από αυτά που παρατηρήθηκαν στην Ευρωζώνη το 2010 όπου οι αυτόματοι σταθεροποιητές έχασαν το λόγο ύπαρξής τους. Μέχρι το 2009 όλοι έλεγαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Ευρωζώνη είναι καλύτερα εξοπλισμένοι από ότι οι Αμερικανοί για αντιμετώπιση κρίσεων. Διότι αυτό ο χώρο διαθέτει του αυτόματους σταθεροποιητέ που είναι ισχυροί. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι από το 2010 και μετά οι διάφορε στατηγικές εξόδου από την κρίση και εξυγίανση δημοσιονομική οδήγησαν σε καταστροφή τη βάση που αντιπροσώπευαν αυτοί οι αυτόματοι σταθεροποιητέ. Άρα μιλούμε για έναν τετραγωνισμό του κύκλου που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να βγούμε από αυτό το δίλημα και το πρόβλημα. Αυτή η πρόταση έχει τεθεί επιτάπητος σαν μια ενδεχόμενη δυνατότητα, σαν μια επιλογή. Δεν είναι η λύση που προτείνεται. Μία από τις λύσεις. Ένα από τα ενδεχόμενα που πρέπει να επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να διερευνήσει δηλαδή τη δυνατότητα μέσω πράσινης βίβλου. Για να διαφωτιστεί η δημόσια συζήτηση. Αντί να αρνείται να εξετάσει την δυσκολία και να επεξεργαστεί βάση προτάσεων που μπορούν να ε, συζητηθούν. Αν υπάρχουν άλλες καλύτερες ε, προτάσεις, εγώ μπορώ να τις δω, να τις εξετάσω, να τις μελετήσω με εξίσου μεγάλη προσοχή. Αλλά είναι μία από τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί. Υπάρχουν και άλλες, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές. Κάθε ένας πρέπει να δει ότι υπό τις παρούς συνθήκες η λειτουργία της Ευρωζώνης δεν είναι βέλτιστη και δεν αρκεί η εξυγίανση και η κάλυψη των ελλημάτων των ελληματικών χωρών για να καλυφθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχουν κοινωνικές συνέπειες, έχουν συνέπειες για τους σταθεροποιητές επίσης, για να γίνει βιώσιμη η Ευρωζώνη. Ζητώ συγγνώμη που χρονοτρίβησα για να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, αλλά από ό,τι κατάλαβα θα γίνει βασικό σημείο των διαπραγματεύσεων για το ψήφισμα και γι' αυτό ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξή μου για την πρόταση και να εκφράσω και τη λύπη μου διότι από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε και άλλα μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση εδώ σήμερα. Θεωρώ ότι είναι το τίμημα του συμβιβασμού, το αποδέχομαι, αλλά παρόλα αυτά ήθελα να πω ότι σκέφτομαι. Σταματάμε εδώ τη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε στη, στη ψηφοφορία. Διαδικαστικό. Πραγματικά διαδικαστικό πρέπει να είναι. Η κυρία Κορνέλησεν Συμφωνώ με τον Τι για το περιεχόμενο, αλλά χρειάζεται ένα ψηφίσμα προς συζήτηση στην Ολομέλεια, είναι κρισίμου σημασία. Είναι πολύ επίμαχη πράγματι η τροπολογία μα 109 και θέλω να την αποσύρω σε αυτή τη φάση. Ευχαριστώ για αυτή τη συνεισφορά στην σημερινή μα επιτυχία, λέει η Πρόεδρος. Στο σημείο 7 λοιπόν έχουμε την ψηφοφορία όσον αφορά το σχέδιο ψηφίσματος που θα πρέπει να υποβληθεί στην Ολομέλεια μετά τη συζήτηση για την προφορική ερώτηση. Κάτι επί το οποίο συμφωνήσαμε σε πρώτερη ψηφοφορία. Προφορική ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβληθεί λοιπόν. Στην παράγραφο 1 έχουμε δύο συμβαστικές. Την Ι ψηφίζουμε υπέρ το, το I δηλαδή λατινικό κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H λατινικό υπέρ θα κάνουμε παλήθευση για το I λατινικό. Tout le monde a pu voter? Ψηφίσατε όλοι. Tout le monde a sa carte? Tout le monde a pu voter? Έχετε όλη κάρτα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ. 17 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Συμβαστική H, τεσσάρων ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, τροπολογία 53, τσάμπαουρι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 54, Heinz Becker υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 56 του ιδίου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 του ιδίου υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 57 ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 29 υπέρ 16 κατά Εγκρίνεται λοιπόν. Παράγραφος 2. Συμβαστική J λατινικό από τρεις ομάδες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά. Τροπολογία 58 των πρασίνων. Με συμπληρώνει την J υπέρ. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται. Επαλήθευση ηλεκτρονική για την 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 20 υπέρ, 25 κατά. Πράγματι απορρίπτεται. Με την παράγραφο 2 πάμε στην τροπολογία 63. Χάινς Μπέκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 από τους πρασίνους υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 65 Heinz Becker υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 65. Τροπολογία 65, πέρας ψηφοφορίας, 22, υπέρ, 23 ψήφοι κατά. Χρειαζόταν αυτός ο έλεγχος, απορρίπτεται. Δεν θα κλάψει ο κ. Μπέκερ, είχε μεγάλες επιτυχίες ήδη. Παράγραφος 3, έχουμε τρεις ψηφ, ε, τροπολογίες διαγραφής υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία κάπα λατινικό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 με προφορική τροπολογία που έγινε δεκτή από την εισηγήτρια υπέρ της τροπολογίας 72 ως ετροποποίηθη κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 5 α περιμένετε ξέχασα να χρησιμοποιήσω τη μηχανή του χρόνου 69 και 70 ήταν συμβατές θα τις ψηφίσουμε λοιπόν 69. Αλεχάνδρο Σέρκα, σαν προσθήκη, υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Τροπολογία 70 των πρασίνων υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Επανερχόμαστε στην παράγραφο 5, τροπολογία 73 για διαγραφή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε λατινικό, δύο ομάδες την παρουσίασαν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος λοιπόν για την τροπολογία τη συμβαστική L λατινικό. Άρχεται η ψηφοφορία. το λίγο. Πέρας. 32 υπέρ, 13 ψήφοι κατά, σαφώς εγκρίνεται. Τροπολογία 78 των πρασίνων υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 79 της ίδιας ομάδας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 τροπολογία 80 για διαγραφή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική M από τέσσερις ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 7 συμβιβαστική N τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με την παράγραφο 7 τροπολογία 87 Heinz Becker υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 8 συμβαστική O από 4 ομάδες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 88 Αλεχάνδρος Σέρκας σαν ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 9 απεσύρθη. Ερχόμαστε μετά την παράγραφο 9. Στην τροπολογία 96 Αλεχάνδρος Σέρκας υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι υπορρίπτεται αλλά θα γίνει επαλήθευση για την 96 λεκτονικό έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται λέει η Πρόεδρος αλλά θα κάνουμε επαλήθευση. Ξεκινάει η ψηφοφορία για την 96. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 37 υπέρ, 8 κατά. Πού είχα τα μάτια μου, σαφώς εγκρίνεται. Τροπολογία 97, Αλεχάνδρος Σέρκας υπέρ, κατά, αποχές, σαφώς απορρίπτεται. Παράγραφος 10, απεσύρθη. Ψηφίζουμε λοιπόν την παράγραφο 11 την τροπολογία διαγραφής 102 και 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 104 Αλεχάνδρος Σέρκας υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 11, την παράγραφο 11 στην αρχή μορφή υπέρ, Α, δεν χρειάζεται. Η παράγραφος 11 Εγκρίθηκε στην αρχική της μορφή, λέει η Πρόεδρος. Παράγραφος 12. Τρεις τροπολογίες διαγραφής 105, 106, 107 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται συμβιβαστική πύλη από το ΕΛΚ σοσιαλιστές και πρασίνους να κάνουμε έλεγχο ότι αυτή η περίπτωση Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι εναντίον. Άρα η συμβαστική καταπίπτει αντίθετα από αυτό που είχαμε συμφωνήσει με το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές και τους πρασίνους εκπλήττομαι από το αποτέλεσμα και εκπλήττομαι που δεν ενημερώθηκα για την θέση, την αλλαγή των θέσεων των πολιτικών κομμάτων πριν την ψηφοφορία. Κοιτάξτε, αν ψηφίσετε τις τροπολογίες διαγραφής για την παράγραφο που υπάρχει συμβαστική, δεν μπορείτε να ψηφίσετε πλέον ε, την συμβαστική. Είναι βασικός κανόνας αυτός. Συγγνώμη, και εμένα με ε, εκπλήσει αυτός ο τρόπος ε, ψηφοφορίας διότι δημιουργεί συγχύσεις. Δηλαδή πρώτα πρέπει να ψηφίζουμε τον συμβασμό. Πρώτα ψηφίζουμε τον συμβασμό και μετά τις τροπολογίες. Αλλά κατά προτεραιότητα ψηφίζουμε τους συμβασμούς. Γιατί διαφορετικά με επέρχεται σύγχυση. Μπορούμε να επαναλάβουν ψηφοφορία για τη συμβαστική, διότι έχουμε ένα λάθος εδώ στον κατάλογο ψηφοφορίας. Πρόεδρε, θα θέλαμε να επαναληφθεί η ψηφοφορία ως προς το συμβασμούς, ως προς τον π, το συμβασμό π. Ε, Εάν πρέπει να επαναλάβω ψηφοφορία, πρέπει να γίνει επί των τροπολογιών 105, 106, 107. Πρόκειται περί διαγραφής που προτείνεται. Επικρατεί κάποια σύγχυση στον κατάλογο ψηφοφοριών και τη σειρά. Με επαναλαμβάνει η γραμματεία ότι ψηφίσαμε τις τροπολογίες διαγραφής, πάντα ψηφίσαμε τις δια... τροπολογίες διαγραφής πριν τη συμβαστική. Αν η πλειοψηφία των ομάδων και οι συντονιστές του ΕΛΚ ζητούν εκ νέου να ψηφίσουμε τις τροπολογίες 105, 106, 107, μπορούμε να το σκεφτούμε. Θα πρέπει τουλάχιστον ο συντονιστή ή συντονιστές, ε, ο συντονιστής του ΕΛΚ να μου το ζητήσει. Πραγματικά λυπάμαι, Πρόεδρε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ακόμα και αν συμβαστική πει συμπεριλαμβάνει την 108 μου, αλλά είμαι στην μειοψηφία της ομάδας μου. Είμαι στην μειοψηφία στην ομάδα μου. Η πλειοψηφία είπε όχι στους αυτόματους σταθεροποιητέ. και είπαν όχι στην πράσινη βίβλο. Δεν το θέλουν αυτό να αναφέρεται στο κείμενο. Λοιπόν, οι 105, 106, 107 θα ψηφίσουμε κατά και ψηφίσαμε κατά και όλα αυτά αντιστοιχούν σε αυτά που λέγαμε μεταξύ μας πριν. Ιδού, αυτό είναι το αποτέλεσμα, συμβαίνει, πρόκειται περί δημοκρατίας, έτσι είναι η δημοκρατία κυρία Πρόεδρε. Να σας ξαναδιαβάσω το κείμενο της συμβαστικής πι, όπως το επεξεργαστήκαμε στη συνεδρίασή μας χτες το βράδυ. Η συμβαστική πι λατινικό λοιπόν που έχετε όλοι στα χέρια σας αντιστοιχεί αγαπητέ Τζαμπάουρη στη βαστική που θέλατε διότι λέει εκφράζεται τη λύπη της για την έλλειψη του ρόλου των σταθεροποιητού στην Αναγκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Δευτέρας Οκτωβρίου του 2013. Το θέμα του αυτόματου χαρακτήρα και της πράσινης βίβλου δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμβαστική πι. Δεν υπάρχει τέτοια αμνία. Θα ήθελα μαζί με τους άλλους συντονιστές να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, διότι είναι παράλογο το ΕΛΚ να δέχεται ένα συμβασμό και τώρα να η θέση διαφέρει από το συμβιβασμό ο οποίος επετεύχθη χτες. Δηλαδή ψηφίσαμε μηχανικά, αλλά όταν το συνειδητοποίησαν κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Πρόκειται για έτοιμα στο οποίο αν δεν αντιτάσσεται κανείς θα ήθελα να ληφθεί υπόψη. Και αυτό είναι υπέρ της δημοκρατίας και όχι κατά. Όσον αφορά εμένα, δεν καταλαβαίνω γιατί 105, 106, 107 θα σκοτώσουν την συμβαστική π. Η συμβαστική π μοιάζει με την 105, 106, 107, δεν ακριβώ ακριβώς ίδια. Πιστεύω ότι αφού ψηφίσαμε την 105, 106, 107, μπορούμε να ψηφίσουμε τη συμβαστική π και μπορούμε να πούμε ναι στη συμβαστική. Υπάρχει αντίδραση στη διαδικασία, στην πρόταση που έκανε ο Τσαμπαωρή. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Λοιπόν, ψηφίζουμε τη συμβαστική π, λατινικό. Η κυρία Σαΐα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ανήκω σε αυτούς που έκανε τροπολογία από αυτές που ψηφίσαμε. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Κάποιοι από εμά θέλουν διαγραφή της παραγράφου 12, εξ διαγραφή. να διαγραφεί. Και αυτό που κάναμε ψηφοφορία είναι ότι κερδίσαμε. Είναι παράξενο λοιπόν τώρα να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Ξε... Κερδίσαν την ψηφοφορία, ήταν πραγματική ψηφοφορία, πραγματική κατάσταση Καμιά φορά το πολιτικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που ικανοποιεί τους πάντες. Ήταν πολιτική ψηφοφορία και πολιτικό το αποτέλεσμα. Ελπίζω λοιπόν που αυτοί που ιτήθηκαν να αποδεχτούν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εγώ δεν θέλω να ξαναρχίσουμε συζήτηση, λέει η Πρόεδρος. Άκουσα την πρόταση του Τσαμπαωρή. Θεωρεί ότι το, ο συμβαστική π που δεν είναι η παράγραφος 12 είναι ένα νέο σημείο που δεν έχει καμία σχέση εν τέλει με το περιεχόμενο της αρχικής παραγράφου 12 που μπορεί να ψηφιστεί ξεχωριστά από την παράγραφο 12. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν, θα ψηφίσουμε ούτως υπέρ της συμβαστικής ποιη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παραγράφο 12, τροπολογία 109, αυτή έχει αποσυρθεί. Παράγραφος 13, τροπολογία 110 της κυρίας Σαρίες Αΐα αφορά διαγραφή που θα κάνει να καταπέσει η συμβαστική Q των, του ΕΛΚ, των σοσιαλιστών, της φιλελευθέρων και των Πασίνων. Ποιος είναι υπέρ της 110. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. Ψηφίζουμε τη συμβαστική Q λατινικό τεσσάρων ομάδων. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13, τροπολογία 112 της κυρίας Ντανούτα Ιασλοβιέσκα. Εδώ έχουμε και προφορική τροπολογία που έγινε δεκτή από την συντάκτια τροπολογίας. Ψηφίζουμε την 112 που τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 13, τροπολογία 113 που υπευλήθη από τους πράσινους που είναι συμβατοί με τη συμβαστική ο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 14. Συμβαστική R λατινικό, ΕΛΚ, σοσιαλιστών, φιλελευθέρων και πρασίνων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 15. Έχουμε, η κυρία Κορνέλησεν. παρατήρησα ότι μετά τη συμβαστική π έχουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας που πρέπει να ψηφιστεί σαν προσθήκη της συμβαστικής π. Επαναλαμβάνει το αίτημα για σταθεροποιητές και την πράσινη βίβλο. Δεν νομίζω ότι το ψηφίσαμε αυτό. Δεν ψηφίσαμε την προστίκη, τη συμπλήρωση. Θεωρήσαμε ότι η 12 είχε διαγραφεί και ότι ψηφίσαμε τη συμβαστική πι σαν κάτι καινούριο, νέο. Δεν μπορούμε να ξανοίξουν τη συζήτηση. Όλοι συμφωνούν με αυτή την ερμηνεία. Τέλεια. Παράγραφος 15 έχουμε δύο τροπολογίες διαγραφής. 116 Σαρία Σαΐα και 117 Φιλίπ Τεμπάκερ. Τροπολογίες διαγραφής. Άρα θα καταπέσει η ΕΣ του ΕΛ, Σοσιαλιστών, Άλντε και Πρασίνων. Ποιο είναι υπέρ των τροπολογιών 116-117. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική S των τεσσάρων προαναφερθήσεων ομάδων. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 15, τροπολογία 119 των Πρασίνων υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 119. Ξεκινάει η ψηφοφορία μας. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 21 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι εναντίον, 4 αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 16. Τροπολογία 120 Σάρια Σαΐα. Περί Αν περάσει δεν ψηφίζουμε την τι. Ποιος είναι υπέρ της 120. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τι τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε σε θεολογικές αναφορές. επτά Έχουν προφορική τροπολογία. Υπάρχουν αντιρρήσεις όσον αφορά την προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχει. Ψηφίζουμε την αιτιολογική αναφορά 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε τροπολογία 1. Αλεχάνδρος Σέρκας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε μετά τη 15, την τελική αναφορά, έχουμε τροπολογία 2 των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά τη λογική αναφορά 15 τροπολογία 3 Αλεχάνδρο Σέρκας υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, τελογική σκέψη D λατινικό συμβαστική α τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τη λογική σκέψη ε, ε, ε τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την έξι τσάμπα ορί. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 20 υπέρ, 25 εναντίον. Δεν εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F, λατινικό, τροπολογία 7 του ιδίου, περί διαγραφής, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη G, τοπολογία 9, Αλεχάνδρος Σέρκας, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8, Τσαμπορί, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μετά την λογική σκέψη G, τροπολογία 10 των πρασίνων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τη λογική σκέψη H, συμβαστική B, τριών ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη I, τοπολογία 13 ορί. διαδιαγραφή υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 13. Ξεκινάει. Ψηφίσατε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 22 υπέρ, 22 κατά, η ισοψηφία δεν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα μετά το Ι, την 14 του Αλεχάνδρου Σέρκα υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίζεται πλέον. Υπέρ 14. Κατά. Επαλήθευση 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι Πέρασε. 25 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. M σε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μετά την, τον συμβιβασμό, μετά το M η 17 καταπίπτει, άρα μετά το M φτάνουμε στη 18 των πρασίνων υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται στο N, 19, σάρια σάρια, και εκπίπτει εκείνη τον ΕΛΚ υπέρ της 19. Πρόκειται για διαγραφή. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την δέλτα τριών ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται στο όμικρον τρεις ε, τροπολογίες διαγραφής 21, 22 και 23. Σάριεσά, Τσαπαωρή και Ντεμπάκερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε, επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 24 υπέρ 20 κατά. Εγκρίνεται. Π. Οι τρεις συντάκτες έχουν υποβάλει τρεις τροπολογίες διαγραφής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε για τις 24, 25, 24, 25 και 26. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Οι 24 έναντι 19 και μία αποχή. Εγκρίνεται. Μετά το Π, τροπολογία 27, Αλεχάνδρο Σέρκας, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 28 του ιδίου, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 29 του ιδίου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο Q έχει αποσυρθεί, άρα ψηφίζουμε το R, την ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά το ε, έχουμε τις 35 και 36 για διαγραφή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Στο τι θέλετε να επαληθεύσουμε, επαληθεύουμε τις 35 και 36. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 24 έναντι ενός. Έχετε δίκιο. Εγκρίνεται. Στο ΤΑΦ 37. Δεμπάκερ. Για διαγραφή και πάλι. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε, γιατί δεν είναι απολύτως ε, σίγουρο το αποτέλεσμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 υπέρ, 20 κατά, μία αποχή, άρα εγκρίνεται. Στο U, τρεις τροπολογίες διαγραφής 38, 39 και 40 για να καταπέσει το F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Άρα καταπίπτει ο συμβασμός F, επαλήθευση, επαλήθευση αν το επιθυμείτε. Η κυρία Σάι είναι σίγουρη ότι κέρδισε, ότι νίκησε. Ας επαληθεύσουμε. 38, 39, 40. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 24 έναντι 21. Πράγματι εγκρίθηκε μετά το... Α, με συγχωρείτε. Μετά το γιου 43 Αλεχάνδρο Σέρκα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 44 Ντεμπάκερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. WG 4 ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το W τροπολογία 47 των πρασίνων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 6, 2 τροπολογίες διαγραφής υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Tout le monde a pu voter. όλοι. Πέρασε. 33 υπέρ, 6 κατά και 6 αποχές. Σας ευχαριστώ πολύ και βασίζομαι στην υποστήριξη των ομάδων έτσι ώστε το θέμα αυτό να ενταχθεί Στι στις συζητήσεις και να ψηφιστεί στην όλο μέλη. Άρα, ας δούμε το σημείο 2 που σχετίζεται με τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Α, έχουμε και άλλες ψηφοφορίες, λέει ο Πρόεδρος. πάμε συγχωρείτε. έχουμε άλλες τρεις ψηφοφορίες, λέει η πρόεδρος. Στο 8 ψηφίζουμε το σχέδιο Μορέν Σαρτιέ για τη χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσορισμένα κράτη-μέλη. Έχουμε νέα τροπολογίες που μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού υπέρ. Κατά Αποχές ε, απορρίπτονται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Η ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 41 υπέρ, 1 κατά, 3 αποχές. Να συγχαρούμε την ε, εισηγητριά μας. Αυτή η γνωμοδότηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον κύριο Γιάνν Όλμπριχτ από την ε, Περιφερειακή Επιτροπή. Εννέα τώρα ψηφίζουμε την έκθεση Edith Bauer για τα μέτρα που διευκολύνουν την ε, άσκηση δικαιωμάτων των εργαζομένων στα πλαίσια της ελεύθερης κυκλοφορίας των ε, εργαζομένων. Στο άρθρο 1 Υπάρχει ο συμβασμός Β τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Παράγραφος 1. B. W. Τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το B. Τροπολογία 13 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 παράγραφος 1 μετά το B, δύο τροπολογίες παρόμοιες 106 και η ΦΑΜ παράγραφος 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Άρθρο 2. Παράγραφος 1. c 108 της Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 2, παράγραφος 1, C, νέο, 109, Τόμας Χέντελ, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες, 21 φαμ και 110, Κορνέλισεν, υπέρ. Ας δούμε καταρχήν την 21 φαμ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110. Κορνέλισεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 2. Παράγραφος 1. D. Εδώ έχουμε δύο τροπολογίες, την 111 Κορνέλισεν και την παράγραφο 22 Φαμ. Τις ψηφίζουμε από εκείνου υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτονται. Επαληθεύουμε λοιπόν. Επαλήθευση. 111 και παράγραφος 22. Υπέρ. Α, ναι. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 25 υπέρ. 20 κατά. Εγκρίνονται οι 112 του Τόμας Χέντελ πίπτη. Α, όχι, είναι συμβατή, είναι συμβατή, άρα ψηφίζουμε. 112 Χέντελ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στο ε τώρα έχουμε την 113 Στάινουρ και Σίπελ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114. Τόμας Χέντελ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.1G. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Άρθρο 2.1. Μετά το G. Ε, y τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά το G117 της Ιούτα Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το G πάλι 118 της Ιδίας και της Σίπελ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Νέα παράγραφος 1, συμβασός α4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και φτάνουμε τώρα στο συμβασμό C, πέντε ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό ζήτα τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κάπα στις ίδιες παραγράφους τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Για το ίδιο άρθρο έχουμε ε, ένα νέο συμβιβασμό τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 3 127. Κορνέλησεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25 φαμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 128 Κορνέλησεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 26 φαμ καταπίπτει, άρα φτάνουμε μετά το ΣΥ Εκατόν τριάντα πέντε Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 Ρέγνερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 133 Μπέκερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 134 Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 136, ψηφίζουμε την 137 Ρέγνε Στάινουρουκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 138 των ιδίων. Και τη ΣΥΠΕΛ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επί του τίτλου ΑΑ υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. ΒΒ πέντε ομάδων υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 144 Κορνέλισεν και Τζιν Λάμπερτ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 145 Κορνέλισεν υπέρ κατά αποχές υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός CC τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στην εισαγωγή 151 Κρίστινσεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δέλτα δέλτα. Τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 φάμ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. 31 φάμ. Ψήφισατε όλοι πέρας. Ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. J. Τριών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 140, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε. Madame Bauer, est 17, Κυρία Μπάουερ, η 17 η δική σας καλύπτεται από το συμβασμό ή όχι. Non. Alors nous pouvons le voter de manière... Όχι, ψηφίζουμε χωριστά. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 155 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 156 δεπάκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32. Φαμ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο συμβιβασμοί. Ε, έψιλον ε, καταρχήν τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το συμβασμό N. Τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 5, παραγραφός 3, νέο α, FF, τεσσάρων πολιτικών ομάδων, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Για τον τίτλο έχουμε δύο παρόμοιες, την 165 Κορνέλισεν και την παράγραφο 33 ΦΑΜ. Υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε. Στον τίτλο, άρθρο 6 τίτλος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 25 υπέρ, 19 κατά, μία αποχή πράγματι εγκρίνεται. Συμβασμός GG τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...169 και παράγραφος 35 φάμ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 171 Κορνέλισεν Λάμπερτ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός HB δύο ομάδων υπέρ κατά αποχές Ας επαληθεύσουμε. HB, επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. 23 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 174, Κορνέλισεν, Λάμπερτ, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. ΦΑΜ 36, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 της εισηγήτριας, υπέρ. Κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Άρθρο 7 παράγραφος 2. Δύο συμβιβασμοί των τεσσάρων ιδίων πολιτικών ομάδων. Η πρώτη είναι η HH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. S ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά το άρθρο 7 παράγραφος 2. Δύο τροπολογίες 183 Κορνέλισεν και παράγραφος 38 ΦΑΜ. ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτονται. Άρθρο 7 παράγραφος 2α 9 184 τροπολογία της ηγήτριας και Μίλαν Κάρμπνοχ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 καταπίπτει, κεφάλαιο 4 νέο, Ψηφίζουμε την τροπολογία 185. Πίρκετ Σίπελ, Γιούτα Steinruck, Evelyn Ρέγνερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 7, νέο, τροπολογία 186 των ιδίων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 187 των ιδίων υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Άρθρο 8, παράγραφος 1, τροπολογία 188, Μαρίγε Κορνέλισεν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άρθρο 8, παράγραφος 2, τροπολογία 189, Γιούτα Στάινρουκ, Πύργη Τσίπελ, Εύλιν Ρέγνερ, υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Επαλήθευση για την 189. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 25 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 190, Μαρία Κορνέλισεν, φαντάζομαι ότι αφορά το άρθρο 8 2 και είναι συμβατή με την τροπολογία 189 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται μετά την παράγραφο 2 το άρθρο 8 τροπολογία 191 Γιούτα Στάινρουκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 10 παράγραφος 1 επαλήθευση για την 191 άρχεται η ψηφοφορία ψηφίσατε όλοι πέρας 20 υπέρ, 21 αντίον. Μηδέν αποχές λέει πρόεδρο, απορρίπτεται. Άρθρο 10, παράγραφος 1, τροπολογία 191, 192, υπέρ. 192, υπέρ. Κατά άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 23, κατά πίπτη, ψηφίζουμε για το άρθρο 10 με την παράγραφο 1, τροπολογία 193, Φιλίπτε Μπάκερ υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Πάντα με την παραγραφό 1, τροπολογία 194, Φιλίπ Πενιού υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 10, παράγραφος 1, δύο τροπολογίες ταυτόσημες, τις ψηφίζουμε μαζί, 195 Φιλίπ Ντεμπάκερ, 196 Φιλ Μπένιον υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε επαλήθευση. Ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 24 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι εναντίον και δύο αποχές σαφώς εγκρίνονται. Αιτιολογική σκέψη 2, συμβιβαστική β, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την τελική σκέψη 3, τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγος 3 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 4. Δύο τροπολογίε, ταυτόσιμε ψηφίζονται. Η 36 της Μαρία Κορνέλισεν και παράγραφος 4 τη επιτροπή Γυναικών. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Μετά την λογική σκέψη 4, τροπολογία 37, επαλήθευση για την 36 και 4 Επιτροπής Γυναικών. Ξεκινάει η ψηφοφορία, ο έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 25 ψήφι υπέρ, 20 ψήφοι εναντίον. Έχετε απόλυτο δίκιο, εγκρίνονται. Μετά την τολική σκέψη 4, την τροπολογία 37, Μαρία Κορνέλισεν, παράγραφο 5 της Επιτροπής Γυναικών. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τελική σκέψη 5, συμβαστική D, 5 ομάδων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 6, συμβαστική ε, 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τη λογική σκέψη 6, συμβαστική τροπολογία 44 των συναδέλφων Ουγγουρεάνου και της ηγητρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 44. Ξεκινάει. Ψηφίσατε όλοι. Ένας σοσιαλίστης παραπάνω. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι εναντίον και δύο αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική σκέψη 8 παράγραφος 7 των γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 47 Μαρία Κορνέλησεν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική σκέψη 9 συμβαστική G 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 10, 51 Μαρία Κορνέλσεν υπέρ, κατά άποχες εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 11, συμβαστική H, 5 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 12, συμβαστική I, 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά σκέψη 12, παράγραφος 8, Επιτροπής Γυναικών υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 13, παράγραφος 9 της Επιτροπής Γυναικών, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 14, τοπολογία 62, Μαρία εν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 14 τροπολογία 63 Μαρίζα Κορνέλισεν, ταυτόσημη με την 10 η Επιτροπή Γυναικών, ψηφίζουμε μαζί υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Τιολογική σκέψη 15, συμβαστική L, 4 ομάδων υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 16, τροπολογία 67, του συναδέλφου Ουγγουρεάνου υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 17, τροπολογία 68, Edith Bauer, Milan, Καμπνοχ, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση για την τροπολογία 68. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά, 4 αποχές. Σαφώς εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 18, δύο τροπολογίες ταυτόσημες, ψηφίζουμε την 69 Edit Bauer και 12 Επιτροπής Γυναικών υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Μετά τελική σκέψη 18, συμβαστική μη 4 ομάδων υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Αριστοτελική σκέψη 18. Τροπολογία 70. Μινοντόρα κλειβέτη υπέρ. Κατά. άποχε. Ε, απορρίπτεται. Αριστοτελική σκέψη 18. Τροπολογία 71. Καταπίπτει. Ψηφίζουμε την τρο... συμβαστική O. Τεσσάρων ομάδων υπέρ. Κατά. απόχε Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 20. Τροπολογία. τεσσάρων ομάδων. Κατά. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 21 Συμβιβαστική Q τεσσάρων ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την λογική σκέψη 21, συμβιβαστική R τριών ομάδων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 22, οι τροπολογίε καταπίπτουν. Μετά τη λογική σκέψη 22 ψηφίζουμε τροπολογία 10 τη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την ελληνική σκέψη 22 πάντα, παράγραφος 14 Επιτροπής Γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη 23, συμβιβαστική U, τεσσάρων ομάδων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά τη λογική σκέψη 24, τροπολογία 96, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τη σκέψη 26, δύο τροπολογίες ταυτόσημες, οι 97 και 17 γυναικών, ψηφίσουμε υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτονται. Αιτιολογική σκέψη 27, τροπολογία 98, Thomas Handel, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Δύο τροπολογίες ταυτόσημες, τι ψηφίζουμε μαζί, τροπολογία 99, Μαρίζη Κονέισεν και παράγραφος 18 Επιτροπής Γυναικών, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, με τελική σκέψη 27, τροπολογία 100, Όλε Κρίστενσεν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο εκθέσεως μέσω ε, ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το τροποποιημένο κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές, 2 ψήφοι εναντίον. Θα ψηφίσουμε την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι εναντίον, 2 αποχές. Ψηφίζουμε τη διαπραγματευτική εντολή. Για να ξεκινήσουν οι πραγματεύσεις, υπενθυμίζω, πρέπει η ειδική πλειοψηφία των μελών που εκπροσωπούν την Επιτροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων να υπερψηφίσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων και αυτή η δική πλειοψηφία στην Επιτροπή μας είναι 26 μέλη. Αν δώσετε την εντολή, η διαπραγματευτική ομάδα θα απαρτίζεται από την πρόεδρό σα την Edith Power, τον κύριο Ole Christensen για τους πρασίνους, ο κύριο Φίλιπ Τεμπάκερ για του Φιλελευθέρου, Μαρίζε Κορνέλισεν για τους πρασίνους, Τόμας Χέντελ για την ΚΟΥΕ και Μίλαν Κράμπνορ για την ECR. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι, πέρας. 40 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος εναντίον, τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας λοιπόν. Και τις ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Πάμε στην τελευταία ψηφοφορία αφορά sur le, le paquet de compromis. Συμβιβαστικό πακέτο. Στις διαπραγματεύσεις για του επομένου νομοθετικού πλαισίου. Για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Η συγγήτριά μας είναι η Μαριάννα Αρκίν. Ψηφίζουμε το κείμενο στο σύνολό του μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου στον τριμερή διάλογο στις 30 Σεπτεμβρίου που επικυρώθηκε από επιστολή της, ε, Κορεπέρ που παρελήφθη στη συνεδρίαση στις 11 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε τη ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 38 ψήφοι υπέρ. 2 ψήφοι εναντίον. 3 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας και σε όλη τη διαπραγματευτική ομάδα. Συνάδελφοι, έχουμε μείνει πίσω μισή ώρα και έχουμε φορτωμένη ημερήσια διατάξη. Παρακαλώ να σταματήσουν οι συζητήσεις. Πρέπει να κάνω σημαντικές, πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. Κάποιες στα αγγλικά, κάποιες γαλλιστή. Πρώτη ανακοίνωση. Ε, για τα Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Ταμεία Επενδύσεων. Στη συνάντηση 11 Σεπτεμβρίου οι συντονιστέ αποφάσισαν να συντάξουν μια γνωμοδότηση για την νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Μακροπρόθεσμα Επενδυτικό Ταμείο για, την, για ε, τις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές ε, επενδύσεις μετά από εξέταση της νομοθετικής πρότασης και της πράσινης φίβλου στην οποία βασίζεται η πρόταση πρωτοβουλία, ο κύριο Γκουτιέρε Πρίο, ο εισηγητής, πρότεινε να μην συνταχθεί γνωμοδότηση στην έκθεση τη Επιτροπή Οικονομικών και Νομικών Υποθέσεων για το σχέδιο κανονισμού, ε, διότι το σχέδιο αυτό αφορά τι ε, νομικές διατάξεις του νέου μέσου και έτσι δεν αφορά άμεσα την Επιτροπή μας. Σύμφωνα με τα όσα ε, διεξήχθησαν στην συνάντηση των συντονιστών, αποφασίσαμε να ανακαλέσουμε την απόφαση που λήφθη 11 Σεπτεμβρίου και να μην συντάξουμε γνωμοδότηση σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Ε, προχωρώντας ταυτόχρονα με τις διαβουλεύσεις για την Πράσινη Βίβλο. Η εξέταση της Πράσινης Βίβλου θα ε, διεξαχθεί αργότερα σήμερα, εάν προλάβουμε. Έπειτα, δεύτερη ανακοίνωση, ε, αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρόγραμμα REFIT. Στην ανακοίνωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεση της να μην προτείνει ένα σύνολο προτάσεων κυρίως την εφαρμογή τη συμφωνία Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τους κομμωτές. Τον ε, καπνό από τα προϊόντα καπνούς, μειοσκελετικές ε, ασθένειες, κάρκινο, γενή ουσίες. Έγινε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων στην τελευταία διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών και η προθεσμία για τις συνεισφορές των Επιτροπών στο τελικό έγγραφο ορίστηκε. Ε, ταυτόχρονα, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων προτίθεται να ε, να αναφερθεί στην ε, ανακοίνωση, στην τελική της ετήσια έκθεση. Η συγητής της Επιτροπής αυτής είναι ο κύριος Καρίμ προθεσμία για τις τροπολογίες που θα περιοριστούν στο πρόγραμμα REFIT θα παραταθεί μέχρι τις 20 ε, Νοεμβρίου το μεσημέρι. Γι' αυτό προθεσμία για τροπολογίες μόνο στην αγγλική γλώσσα για την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και μόνο για το ε, κομμάτι που αφορά το πρόγραμμα REFIT έχει τεθεί για την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα ψηφίσουμε στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης στις 25 ναι. και 26 Νοεμβρίου. 13, όχι 30 Νοεμβρίου, μας συγχωρείτε. Και με τον τρόπο αυτό θα προλάβουμε να υποβάλουμε τις δικές μας τροπολογίες στην έκθεση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Αναμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας. Τρίτη ανακοίνωση. Λοιπόν, αφορά την νομοθεσία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στη συνεδρίαση την έκτακτη της, επί, της στην ψηφοφορία για τη θέση μας, την τελική μας θέση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αυτή θα λάβει χώρα σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας που θα λάβει χώρα στο Στρασβούργο Δευτέρα 18 Νοεμβρίου από τις 7 μέχρι 8.30 για να επικυρωθεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο επ' αυτού. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονισμού και συμφωνία, στη συμφωνία με τη Συγήτρια, θα καταθέσουμε στην Ολομέλεια ονόματι τη Επιτροπή Απασχόληση στην τροπολογία που θετήθηκε στι 9 Ιουλίου, που έχει σαν στόχο την επανεισεγωγή το τμήμα του Κοινωνικού Ταμείου, το 25% τη πολιτική συνοχή δηλαδή. Η συμφωνία που επιτέθη αντιμετωπιστική ομάδα και το Συμβούλιο απερίφθη στην Επιτροπή Απασχόληση με 32 ψήφου υπέρ 32 με 12 για την τροπολογία του 23,25%. Άλλη έκτακτη σύνοδος της Επιτροπής Απασχόλησης, κοινή με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, θα λάβει χώρα στις 21 Νοεμβρίου από τις 8 και 4 μέχρι τις 10, ούτως ώστε να ακουστεί η παρουσίαση πλευράς των Επιτρόπων Άντορ και Ρεν, τις τελευταίες αιτήσεις εξέτασης ανάπτυξης αυτής της θητείας. Βασίζομαι στην παρουσία σας σε αυτές τις δύο συνεδριάσεις, τις έκτακτες συνεδριάσεις. Τέταρτη ανακοίνωση. Ξαναπάω αγγλικά. Αποτελέσματα της άτυπης επίσκεψης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 7 Οκτωβρίου. Η αποστολή αυτή της Επιτροπής Απασχόλησης από το λίγο από εμένα, τον ε, κύριο Κόφ, την κυρία Γιασλοβιέτσκα. Από αυτούς τους τρεις, λοιπόν, ευρωβουλευτές. Από τον κύριο Πάπαδοπούλου επίσης και τον κύριο Άρντεν για τους σοσιαλιστές και από τον κύριο Άλεν από την ομάδα EFD. Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα. Οι τελευταίε εξελίξει στον χρηματοπιστωτικό και οικονομικό τομέα, οι κοινωνικές και πολιτικέ πτυχέ ε, του πλαισίου οικονομική διακυβέρνησης, η, η κατάσταση των ε, της Τραπεζικής Ένωσης, η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων σε πιστώσεις, και η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση και οι μελλοντικές προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα προγράμματα στήριξης. Η συνεδρίαση αυτή ήταν και κλεισμένων των θυρών και δεν θα υπάρξει περαιτέρω σύνοψη των διεργασιών της συνεδρίασης αυτής. Επιπλέον, μια ανακοίνωση σχετικά με την ίδια κοινοβουλευτική συνεδρίαση, άρθρο 13, για το δημοσιονομικό πακέτο που ε, έλαβε χώρα στο Βίλνιους από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Ο συνάδελφό μας Όλε Κρίστενσεν θα μας παρουσιάσει στην επόμενη συνεδρίαση η οποία θα γίνει επίσης στο Βίλνιους. Τα αποτελέσματα θα είναι μια συνεδρίαση ανάμεσα σε μια επιτροπή που ασχολείται σε εθνικό επίπεδο, επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων με τα θέματα της Επιτροπής Απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Βίλνιους, θα πρέπει φυσικά να ασχοληθούμε και με την ε, γενικότερη τη γενικότερη κατάσταση. Επίσης, η κατάσταση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Διεξήχθη μια συνεδρίαση στο Βίλνιους, όπως είπα, από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε στείλει μια αντιπροσωπεία με 8 μέλη. 8 μέλη από τα 16 που είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε. Τα μέλη ήταν τα εξής. Από τις επιτροπές ε, Econ, Empl και budget. Εγώ προσωπικά συμμετείχα εκ μέρους της Επιτροπής αυτής, της Επιτροπής Απασχόλησης. Τώρα δεν θα επεκταθώ, δεν θα αναφερθώ στα εύκολα, θα ήθελα όμως να αναφερθώ στο πιο αμφιλεγόμενο σημείο και συνάμα μια μεγάλη επιτυχία, ένα δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια του Fiscal Compact. Καταρχάς, το ε, πλέον αμφιλεγόμενο σημείο ήταν η διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει εκ των προτέρων ότι αντίθετα ε, με τις επιθυμίες της Προεδρίας ήταν αρκετά ε, νωρί για να συζητήσουμε πάνω στον κανονισμό λειτουργία. Συμφωνήσαμε ότι η ομάδα εργασία που θα αποτελείται από εκπρόσωπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων θα εργαζόταν για ε, να συντάξει ένα προσχέδιο των, ε, του κανονισμού λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Fiscal Compact στο αποτέλεσμα της συνάντησης που έγινε στην Λευκοσία. στην οποία συνάντηση μας εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επίσης μετά από την επιστολή που μας έστειλε το Λιθουανικό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα για το Κοινοβούλιο είναι ένα κρεμές ζήτημα διότι εμεί δεν είχαμε συνεισφέρει μέχρι τώρα μετροπολίτες και τώρα πρέπει να αρχίσουμε τη διαδικασία από την αρχή. Τώρα, όσον αφορά το σχέδιο συμπεράσματο Το Λιθουανικό Κοινοβούλιο μας υπέβαλε ένα σχέδιο μία εβδομάδα πριν τη συνεδρίαση και εμείς η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείναμε να, ε, να δοθεί διαφορετική ονομασία η οποία διέφερε αρκετά από την προηγούμενη. Μετά από συζητήσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες ψηφίστηκε ένα κείμενο στην ολομέλεια που ακολούθησε. Το Λιθουανικό Κοινοβούλιο μεταβίβασε και αυτό με τη σειρά του τα αποτελέσματα και μπορώ να πω ότι η Λιθουανική Προεδρία έλαβε υπόψη της ε, πολλά από τα σημεία που είχαν δημοσιευτεί στην κοινή δήλωση. Ο τίτλος τώρα του συνεδρίου. Να πω εδώ τα εξής. Το Λιθουανικό Κοινοβούλιο είχε υποβάλει ε, όλες τις λεπτομέρειες για το συνέδριο υπό τον τίτλο «Διακοινοβουλευτική συνεδρίαση για την διακυβερνητική και οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη». Αυτό αντιτίθεται σε όλο το σκεπτικό του άρθρου 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου, διότι όπως γνωρίζετε αυτό το σύμφωνο αναφέρεται στην δημοσιονομική πολιτική και εάν τώρα διεξάγεται μια συνεδρίαση για χρηματοοικονομικά θέματα τα οποία βρίσκονται στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, το ζήτημα περιπλέκεται και γίνεται κάπως περίεργο. Δεν ε, στάθηκε δυνατόν να αλλάξουμε τον τίτλο κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας, όμως κατέστη σαφές στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου από τη Λιθουανική Προεδρία ότι το θέμα αυτό θα μεταφερθεί στην επόμενη, στην Ελληνική Προεδρία, η οποία θα έχει και το έργο της επίλυσης του προβλήματος. Αυτά για αυτό το θέμα. Τώρα θα διοργανωθεί μαζί με το Κοινοβούλιο και την Ελληνική Προεδρία η δεύτερη σχετική συνεδρίαση τον Ιανουάριο του 2014 και οι συντονιστές έχουν ήδη ενημερωθεί για τις προτάσεις επί του περιεχομένου της συνεδρίασης αυτής. και έχουμε ήδη συζητήσει μαζί του για τις εξελίξεις. Αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω. Αυτό το συνέδριο προστίθεται σε μία σειρά ε, άλλων συνεδρίων. Καταρχάς το συνέδριο και έπειτα το συνέδριο που ε, θα αφορά την εξωτερική πολιτική. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ε, είμαστε λεπτομερής και άκριβης σχετικά με, με το περιεχόμενο και να αποφύγουμε τις αλληλοεπικαλύψεις. Εγώ πιστεύω λοιπόν πως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό αυτό το άρθρο 13, συνεδρίες του άρθρου 13 να παραμείνει υπό το δημοσιονομικό σύμφωνο, το οποίο αφορά δημοσιονομικά ζητήματα. Και ένα θέμα προς διαβούλευση Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων. Έκτον, δεν έγινε καμία ακύρωση διερμηνίας, αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο και έβδομο να σας πω ότι ο φάκελος των συνεδριάσεων είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονικά ε, με βάση την εφαρμογή e-meeting. Και ε, έχετε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία επιγραμμικά. Έχετε παρατηρήσεις όχι, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και τώρα περνάμε στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης και δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας, ε, Ρία Όμιν Ρόιτεν, για να μας πει πώς είχαν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τη δυνατότητα μεταφοράς των ε, συμπληρωματικών συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Ε, collega's, we hopen dat we morgen de onderhandeling kunnen afsluiten. Ελπίζω αύριο να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις και αυτό είναι το καλό κομμάτι. Δεν ξέρουμε όμως αν θα τα καταφέρουμε. Διότι και οι πρέσβεις θα διαπραγματευτούν αύριο για το σημείο αυτό. Πριν 10 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε υποβληθεί μια πρόταση σχετικά με την δυνατότητα που θα έπρεπε να είχαν οι άνθρωποι να μεταφέρουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα από το ένα κράτος στο άλλο. Αυτή η πρόταση έχει αλλάξει ριζικά. Τώρα πρόκειται για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και η νέα οδηγία λέει ότι μετά από μία περίοδο τριών ετών έχει κάποιος το δικαίωμα να πάρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα από τη μία χώρα και να τα μεταφέρει σε άλλη. Και αυτή η περίοδος των τριών ετών είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα τρία χρόνια δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο σε αυτό το ζήτημα. Έπειτα, η οδηγία αυτή ισχύει μόνο για όσους εργάστηκαν σε διασυνοριακή, διασυνοριακές συνθήκες απασχόλησης. Μόνο σε εκείνους, όχι σε απασχολούμενους που εργάστηκαν σε ένα κράτος μέλος. Γι' αυτό εμεί ζητούμε να Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιτρέψει την μεταφορά των συνταξιοδοτικών ε, δικαιωμάτων, όχι μόνο σε όσους εργάστηκαν ε, διασυνοριακά, αλλά και στους υπόλοιπους. Δύο χώρες ε, διατύπωσαν τις αντιρρήσεις τους, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία, για αυτήν την τροποποίηση. Έπειτα, τι γίνεται με τους εργαζόμενους οι οποίοι μετακομίζουν και ξαφνικά γίνονται διασυνοριακοί εργαζόμενοι. Καταρχάς, να σας μιλήσω ειλικρινά. Δεν είδα το, το παραθυράκι εδώ, το κόλπο αν θέλετε. Πολλοί συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε ένα νομικό παραθυράκι και θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, ζω στο Βέλγιο και μετακομίζω στο Λουξεμβούργο, ας πούμε. Και μετά, επί τρία χρόνια, θα έχω συνταξιοδοτικά δικαιώματα βασισμένα σε αυτά που θα έχω δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών. θα χαρακτηρίζεται κάποιος ε, ως διασυνοριακός εργαζόμενος, όχι μόνο ένα έχει εργαστεί για τρία χρόνια, εάν έχει μετακομίσει σε άλλο κράτος μέλος, όχι απαραίτητα σε άλλη εταιρεία και μετά από δύο χρόνια επιστρέψει στη χώρα του. Ας φανταστούμε τώρα ότι όταν, είμαι, όταν γίνω 65, ως τελευταίο στάδιο της ε, καριέρας μου, μετακομίσω στη Γερμανία και εργαστώ εκεί για τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό. Θα πληρώ τις προϋποθέσεις της οδηγίας, όμως όχι τις προϋποθέσεις ενός εξωτερικού απασχολούμενου. Θα θέλω λοιπόν να, να συνταξιοδοτηθώ στα 68, δεν θα έχω όμως το δικαίωμα αυτό. Το επιχείρημα αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα σωστό και εμείς θεωρούμε ότι η οδηγία αυτή έχει πολλές αμφισημίες. Αυτά λοιπόν σε γενικές γραμμές είναι τα πιο σημαντικά σημεία. Τόμας Μάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ρία, για την έκθεση. Ήθελα όμως μερικές διευκρινήσεις. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει το θέμα, έχουμε συμφωνήσει ότι διαφωνούμε και... Και αναφέρθηκε σε ότι δύο, δύο κράτη-μέλη έχουν πρόβλημα με αυτό. Εγώ νομίζω πως είναι περισσότερα. Έχουμε μία ρύθμιση η οποία αφορά μόνο τις διασυνοριακές περιπτώσεις, όταν κάποιος δηλαδή μένει σε μια χώρα και εργάζεται σε μια άλλη. Τώρα, αυτό που, αυτή η προσπάθεια που παρατηρείται είναι να ε, αφορά όχι μόνο ε, δύο κρατημέλη, αλλά να αφορά και τους εργαζόμενους στο ίδιο, σε ένα κράτος μέλος. Αν μπορούσες να μου το εξηγήσει, θα το εκτιμούσα στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στον, ε, στο θέμα αυτό, αλλά όχι μόνο εκεί. Θα ήταν λοιπόν καλό εάν μας επαναλάμβανες και μας εξηγούσες. Έπειτα, όσον αφορά την προθεσμία των ε, τριών ετών, ξέρω ότι χρειάζεται να μειωθεί αυτή η προθεσμία. Όμως ε, πραγματικά αυτά είναι τα κατώτατα όρια που μπορούμε να θέσουμε τα τρία χρόνια πρέπει να είναι σίγουρα. Δεν καταλαβαίνω τη στάση σου. Τη βρίσκω άκαπτη. Έπειτα, όσον αφορά την ε, συντόμευση από πέντε σε τρία χρόνια της ε, προθεσμίας εφαρμογής. Ε, θα ήθελα εδώ να τοποθετηθείς, γιατί δεν το έχεις κάνει. Και έπειτα, αναφέρεσαι σε αυτή την οδηγία η οποία καλύπτει ένα εύρος δυνατοτήτων και αναφέρεσαι σε κάποια παραθυράκια σε αυτή την οδηγία. Και θα ήθελες να ασχοληθούμε με αυτά. Και πιστεύω πως αυτό πρέπει να το κάνουμε και αν το κάνουμε σωστά θα έχουμε ένα πλεονέκτημα σε μελλοντικό τριμερή διάλογο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ξέρεις ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις και τις έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια και να σου πω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν και ομάδες εργασίας οι οποίες ε, εργάζονται με τελείως διαφορετικές συνθήκες για, τα τελείως, για τελείως διαφορετικά, διαφορετικούς στόχους αυτό που χρειαζόμαστε είναι ενδελέχεια. Πρέπει οι διαπραγματευτικές ομάδες να έχουν μία ενιαία θέση, όπως το Συμβούλιο έτσι και εμείς, και χρειάζεται γι' αυτό πολύ καλή ενημέρωση. Όμως, ε, όπως και να έχει, χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρθηκε σε στην διαφάνεια και πιστεύω πως είσαι αρμόδια για το θέμα αυτό. Ja słusznie zwróciłaś uwagę, że tak naprawdę diabeł Ευχαριστώ πολύ. Όντω, οι λεπτομέρειε είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ρωτήσω ποιο το επιχείρημα για, τα, για το ελάχιστο των τριών ετών. Συνολικά τρία συνεχόμενα χρόνια ή τρία χρόνια καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου κάποιου ανθρώπου. Πώς ακριβώς ορίζονται τα τρία χρόνια. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Θα ήθελα να πω ότι στις συζητήσεις με το Συμβούλιο υπάρχει διαφωνία επί της ουσίας για το αντικείμενο αυτού του νομοθετήματος και αν ξεμπλοκαριστούν οι διαπραγματεύσεις, αν έγινε αυτό στο Συμβούλιο, είναι διότι υπάρχει μια κινητικότητα ενώ κατά την άποψη του Κοινοβουλίου το θέμα της ισότητας των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να παραμερίσουμε ακόμα και όταν υπάρχει ενισχυμένη κινητικότητα όπως ε, ζήτησε το Συμβούλιο και ιδιαίτερα ορισμένα μέλη του Συμβουλίου. Αλλά υπάρχει διαφωνία επί του ουσίας, ε, ελπίζω όμως αυτό να μην προδικάσει τις συζητήσεις η εισηγήτρια και την κατάληξη των συζητήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα απαντήσω σύντομα στην Τανούτα και στον Τόμας. Ε, το Συμβούλιο πρότεινε, επαναλαμβάνω, ότι ο χρόνος αναμονής μέχρι κάποιος να έχει δικαίωμα σύνταξης θα είναι τα τρία χρόνια. Αυτό, Τανούτα σημαίνει ότι σε αυτά τα τρία χρόνια κάποιος πρέπει να εργάζεται. Κατάλαβες. Πρέπει κάποιος επί τρία χρόνια να έχει εργαστεί για κάποιον εργοδότη μόνο τότε. Και αυτό είναι ο ελάχιστο ε, χρόνος. Μόνο τότε μπορεί να έχει κάποιος ε, δικαίωμα για σύνταξη. Έπειτα, κυρία Πρόεδρε, Άκουσα και τον ε, Τόμας που το ανέφερε και έχω απαντήσει και σε πολλές επιστολές γερμανικών ενώσεων. Εμείς προσπαθούμε, είναι και στόχος μας, να δημιουργήσουμε μια σωστή νομική βάση. Εάν κάποιος ε, θέλει να μετακομίσει σε μια άλλη χώρα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να το κάνει χωρίς να δημιουργεί αυτό προβλήματα έπειτα. Και εμείς επιμείναμε με γραπτή επιστολή μας ότι αυτά που ισχύουν τώρα για τη διασυνοριακή εργασία πρέπει να εφαρμοστούν και στη Γερμανία και στο Λουξεμβούργο. Εσείς οι δύο είστε οι μόνες χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζετε αυτές τις διατάξεις. Αυτό που δεν θέλω σε καμία περίπτωση είναι εάν κάποιος εργαζόμενος, έχει αποκτήσει δικαίωμα για σύνταξη μετά από τρία χρόνια, να χάσει το δικαίωμα αυτό επειδή δεν επιστρέφει στη χώρα στην οποία το απέκτησε. Αυτό είναι ένας ε, πολύ σοβαρός ε, περιορισμός και αυτό θέλουμε να το αποτρέψουμε οπωσδήποτε. Ε, Θα έχουμε τη δυνατότητα να επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση μετά τον επόμενο τριμερή διάλογο. Θα λάβει χώρα αύριο. Και θα δούμε αν θα καταλήξει κάπου ή όχι. Και σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία αύριο. Χωρίς να χαθούν τα ουσιώδη όμως. Στο σημείο 13 ερχόμαστε στην έκθεση Γιούτα Στάινρουκ θα εξετάσουμε τις τροπολογίες της εκθέσεως πρωτοβουλίας της. Αφορά σωματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη. 121 τροπολογίες κατετέθησαν. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι εργάστηκαν εντατικά για την έκθεση αυτή. Τώρα μια γενική επισκόπηση των τροπολογιών. Ασχολούμαστε με τις νέες προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με τα νέα δεδομένα που έχουμε, με τις επιθεωρήσεις εργασίας. Οι τροπολογίες αφορούν ε, τομείς ε, ασφάλειας και υγείας, ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Ορισμένες τροπολογίες αφορούν ε, την, τους αυτοαπασχολούμενους. Άλλες τροπολογίες αναφέρονται στην κατάρτιση, στον ρόλο των πληροφοριοδοτών και την προστασία τους. Αναφέρεται επίσης ε, η επιθυμία για εντονότερες ε, κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων. Αναφέρεται η ε, απόσπαση των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους, η συμπερίληψη των συνδικάτων στις επιθεωρήσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο δεν συμφωνούν όλοι. Όμως ε, από τις σκανδιναβικές χώρες έχουμε πάρα πολύ καλές εμπειρίες σχετικά με την συμπερίληψη των συνδικάτων σε αποθεωρήσεις εργασίας. Επίσης, ε, επιθεωρήσεις εργασίας στους κατοίκων εργαζόμενους. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς συναδέλφους είναι οι επιθεωρήσεις για μετακινούμενους εργαζόμενους. Ε, θεωρώ ότι ορισμένες τροπολογίες αποδυναμώνουν την αρχική πρόταση. Τώρα υπάρχουν επίσης τροπολογίες οι οποίες ε, έχουν νέες προτάσεις, κ. Μπουλάν για παράδειγμα, ο οποίος ε, ζητεί μία υποχρεωτική ιατρική εξέταση, η επίσης τροπολογία του κυρίου Σαρία για τις ε, δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες πρέπει να ε, αποστέλλονται άμεσα στις ε, αρχές επιθεώρησης εργασίας. Επίσης ε, αναφέρεται σε τροπολογίες η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής των πρακτικών και συνεργασίας που επιθυμούμε να συσταθεί στα πλαίσια της ε, Eurofund. Θεωρώ πως οι γενικές γραμμές η συνεργασία ήταν ε, πολύ καλή, δεν είχαμε πρόβλημα σε, για να οδηγηθούμε σε κάποιον συμβιβασμό. Αύριο θα συζητήσουμε και μεθαύριο την Πέμπτη θα έχουμε την πρώτη συνάντηση. Τώρα οι μεγάλες διαφωνίες ε, εστιάζονται στις ε, πολιτικές, ε, στην πολιτική διάσταση, ιδιαίτερα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης, Κοινωνικής Ασφάλισης. Μια έχουμε μια πλειοψηφία που επιθυμεί να μην ενισχυθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή διάσταση ελέγχου και αυτό το βρίσκω λυπηρό. διότι έχουμε πολλά παραδείγματα όχι βέλτιστων αλλά χείριστων πρακτικών και εδώ έχουμε παρατηρήσει ότι και τα κρατημέλη και οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο φόρτο εργασίας σχετικά με τις επιθεωρήσεις εργασίας. Πολλά κρατημέλη αδυνατούν λοιπόν να διεξάγουν εξονυχιστικούς και κατάλληλους έστω ελέγχους ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, τους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Έχουμε πολλές αναφορές από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Κύπρος που μας λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μπορέσουν να ελέγξουν όλες τις περιπτώσεις. Έπειτα, πολλοί συνάδελφοι πρότειναν την, ε, και στήριξαν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας που θα ενισχύσει την ε, επιθεώρηση εργασίας. Επίσης υπάρχουν πολλές τροπολογίες που ζητούν την, ε, την πρόληψη του κοινωνικού ντάμπινγκ, την αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ και υποστηρίζουν πως αυτό θα είναι δυνατόν μέσω αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής που έχουν προτείνει να δημιουργηθεί. Ελπίζω και είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε σε συμβιβασμό τουλάχιστον στα σημαντικότερα θέματα και θα ήθελα σε αυτό το σημείο κλείνοντα να ευχαριστήσω ξανά όλους τους κοιόδης εισηγητές. Καλώς, Φιλίππουλου, πρώτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να ευχαριστήσω την Γιούτα για τη δουλειά που έκανε να της πω ότι περιμένω τις συμβαστικές τροπολογίες που προτείνει, αλλά πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε σε πάρα πολλά σημεία. Κατέθεσα 17 τροπολογίες εγώ ίδιος, χωρίς να επαναλάβω τα υποθέντα, οι τροπολογίες επί των οποίων ήθελα να προχωρήσουμε αφορά τις επιθεωρήσεις στην περίπτωση απόσπασης εργαζομένων και επιθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις να προβλέπεται η αύξηση των επιθεωρήσεων επί μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πολύ μικρών εργοταξίων, να μην καταφέρουμε να σταματήσει, ε, να... Να, να εκμεταλλεύονται την έλλειψη ενημέρωσης των εργαζομένων. Χρειάζεται ενημέρωση και επίσης και το θέμα της ε, περίθαλψης θα πρέπει ε, οι ξένες γλώσσες να λαμβάνονται υπόψη στον αφορά την εκπαίδευση των δεχτών και κοινωνικέ θα πρέπει επίσης να, φεύγει, να φεύγει η ετικέτα η έγκριση ενός, να θεωρείται κάποια ευρωπαϊκή εταιρεία ότι είναι ευρωπαϊκή συμμορφότητα, ευρωπαϊκή νομοθεσία αν δεν πληρεί αυτούς τους κανόνες. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται και η Euroform, η πλατφόρμα αυτή, ούτως ώστε να υπάρχει μια βάση το Ίδρυμα χρησιμοποιείται για να μπορεί να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους επιθεωρητές εργασίας. Χρειάζεται η συνολική συνεργασία και έτσι μπορεί να καταπονηθεί και η παράνομη παροχή υπηρεσιών. Σε μια τη τροπολογία υπάρχει μια πρόταση ώστε να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρό σε πολλέ γλώσσε, χωρί να περιορίζεται το επίπεδο της μετάφρασης ε, λόγω με μακροσκελών εγγράφων, του μεγέθους των εγγράφων, αλλά πρέπει συστηματικά να γίνεται μετάφραση. Αυτό όσον αφορά ε, τα συμπληρωματικά σημεία που ήθελα να αναφέρω, σημεία που δεν ανακοινώθηκαν από τη Γιούτα, αλλά εν γέννη νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και θέλω να συγχαρώ τη Γιούτα και περιμένω ανυπόμονα τις ε, συμβαστικές ε, τροπολογίες που θα μας προτείνει. Ευχαριστώ. Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, την κυρία Στάινρουκ. Έχω κάποια σχόλια όσον αφορά ε, τα προτινόμενα και προτείνω κάποιες τροποποίησεις που εμείς οι οικολόγοι θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να γίνουν στον αφορά την έκθεση. Καταρχάς πιστεύω ότι ο γενικός τόνος του κειμένου είναι καλός διότι εν γέννη ε, βασιζόμαστε στις ε, αναλύσεις και τα αιτήματα το κείμενο εστιάζεται πολύ σωστά επί του κοινωνικού ντάμπινγκ, από αυτής τη πτυχής είναι κάτι καλό, διότι ξέρουμε ότι το κοινωνικό dumping σήμερα όλο και περισσότερο περνά μέσω της αποσπα... των αποσπασμένων εργαζομένων και είναι καταστροφικό αυτό και είναι καταστροφικό για τα άτομα που ξέρουμε ότι αυτό θα μεταφραστεί με κάποιο τρόπο. Τα άτομα είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης, σκανδαλώδους εκμετάλλευσης, χαμηλή αμοιβή, τα δικαιώματά τους θα στερούνται, προσωπικότητα προσβάλλεται, εξωπρέπεια κλπ. και για την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασία. Κάθε χρόνο 168.000 Ευρωπαίοι πολίτε πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατυχήματα και από ασθένειε που σχετίζονται με την εργασία. Και 7 εκατομμύρια τραυματίζονται σε διάφορα ατυχήματα. Είναι και μια καταστροφή για τι επιχειρήσει. Γιατί? Διότι εάν αυτή δεν κάνει κάποια κόπα, χάνει λοιπόν χάνει τη θέση την ανταγωνιστική και δημιουργεί και προβλήματα ε, από προβλήματα από απώλεια φόρων τα κράτη και τελικά και τα κράτη-μέλη χάνουν την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη μα υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Όταν θέλουμε να ασχοληθούμε λοιπόν το μέλλον τη επιθεώρηση εργασία στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να ρισμονούμε και διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα η έλεγχη από πλευρά επιθεωρητών των κανόνων, από πλευρά επιθεωρητών εργασία. Πρέπει να είναι όμω ομοιόμορφη η εφαρμογή. Αν όλε οι επιχειρήσει, αν όλοι οι εργαζόμενοι, ε, όλοι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσει πρέπει να ελέγχονται. Μετά το κοινωνικό dumping, άλλη πτυχή. Το κοινωνικό dumping δεν περνά μόνο από την ψευδή απόσπαση εργαζομένων. Καμιά φορά γίνονται σεβαστοί κανόνε. Και υπάρχουν και περιπτώσει πραγματικού dumping. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη της εφαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εργασία, ε, μελάχιστος μισθός, έλλειψη διάκρισης, δικαίωμα να νίκει κανείς σε συνδικάτο κλπ. Ε, τρίτη πρόταση μετά, ε, μια αποτελεσματική επιθεώρηση εργασίας είναι μια επιθεώρηση εργασίας που είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι όσον αφορά την υγεία στην εργασία, χρειάζεται να υπάρχουν γνώση την υγεία, να μόνο επαγγελματίε θα μπορούν να τοποθετούνται θεμάτων υγεία, που θα είναι ανεξάρτητοι ειδικοί για θέματα υγεία που θα δημιουργούν αυτού του έλεγχου για την υγεία. Αποτελεσματική επιθεώρηση εργασία τι είναι. Επιθεώρηση εργασία που ωφελείται από ανθρώπινους πόρους σωστού και σωστά επαρκή κονδύλια για να μπορεί να εκτελεί την αποστολή τη. Ιδού εν ολίγηση προσανατολισμοί που θέλω να ακολουθήσω και θα ήθελα να συμπεριλαμβάνω την έκθεσή σας λοιπόν, συγγνώμη διότι στην πρώτη μας συνάντηση δεν θα μπορώ να είμαι παρούσα αλλά πολύ προσεκτικά παρακολουθώ την έκθεσή σας διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ντανούτα Γιασλοβιέσκα και μετά ο συνέφος Κασίν. Ευχαριστώ. Ε, συνάδελφοι, όλοι συμφωνούμε ότι η επιθεώρηση της εργασίας ε, ε, αποτελεί σημαντικό μέρος της καταπολέμησης των καταχρήσεων. Οι επιθεωρήσεις είναι απόλυτα αναγκαίες και δεν μπορούν να αποτελέσουν μέσω προστατευτισμού. Δηλαδή, μπορούν να βαρύνουν τους εργοδότες και τις εθνικές ε, διοικήσεις. Η έκθεση ε, προβάλλει ιδέες ε, που θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις επιθεωρήσεις και να επιβαρύνουν και τους εργαζόμενους. Δηλαδή μιλάμε για τις εθνικές επιθεωρήσεις που θα πρέπει να περάσουν σε ε, κοινοτικό επίπεδο με τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού φορέα με ένα σύστημα, μια βάση δεδομένων καθώς και ερωτηματολόγια. Αυτό αφορά τις εθνικές αρχές γιατί ξέρουν καλύτερα πώς μπορούν να προβούν σε αυτές τις επιθεωρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλά ε, ερωτηματολόγια τύπου Α1 έχουν ε, εκδοθεί. Θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών να ε, προωθήσουμε την ανταλλαγή δεδομένων και την καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων. Γίνονται πολλές παραβιάσεις του νόμου, ε, κατά συρροή παραβιάσεις, γιατί δεν υπάρχει σωστή ε, γνώση του αντικειμένου από τους εργαζόμενους. Γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τις διασυνοριακές επιθεωρήσεις και η Επιτροπή θα πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις στους εργοδότες. Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπερβολικός παρεμβατισμός στα, στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Θα πρέπει να υποστηρίξει η Επιτροπή τις εθνικές αρχές σε αυτή τη διαδικασία κατάρτισης. Επίσης, μιλάμε ε, και για την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ε, ε, εργαζόμαστε επί της οδηγίας και αναμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο να αναφερθώ και στο σημείο 8 όπου το βελικό σύστημα θεωρείται ένα καλό σύστημα λειτουργίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι το σύστημα αυτό δεν συμβαδίζει με την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό θα πρέπει να απαλληφθεί αυτή η μία στην ε, έκθεση. Δεν θέλουμε πλέον προσκόμματα στην ε, πρόσβαση στην αγορά κατά το δυνατόν. Ως προς τους αποσπασμένους εργαζόμενους πολλές φορές είναι όμοιροι της ε, κατάστασης και θα ήθελα να, να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν υπάρχει αυτή η ομοιρία των εργαζομένων, ναι ή όχι. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Γιούτα, συνάδελφοι, όπως είπα νωρίτερα, εκ μέρους της Άλτε πιστεύω πως ε, η έκθεση αυτή θα είναι μια πολύτιμη συνεισφορά όχι μόνο για τις συνθήκες εργασία στην Ευρώπη αλλά και για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι επιθεωρήσεις εργασίας είναι προβληματικές σε πολλά κράτη-μέλη και πολλές φορές ε, από, ε, έχουν προβλήματα έλλειψης ε, πόρων, έλλειψης ε, ανθρώπινου δυναμικού και ελλειπούς εφαρμογής του νόμου. Ορισμένες από τις τροπολογίες μας ίσως φανεί ότι προσπαθούν να περιορίσουν το πεδίο εφαρμογής. Ωστόσο, εμείς στηρίζουμε απόλυτα όλες τις ουσιαστικές και πρακτικές επιτυχίες της πρότασης, διότι πιστεύουμε ότι τα προβλήματα αυτά μπορούν να επιληθούν εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή μας ε, θα μπορέσει να ε, συνεισφέρει σε αυτό. Για παράδειγμα, πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες εργασίας, όμως δεν είναι η δική μας αρμοδιότητα να αναφέρουμε παραβιάσεις. Εμείς έχουμε τροποποιήσει την πρόταση με τις τροπολογίες μας έτσι ώστε να ε, συμφωνεί και με τις άλλες σχετικές προτάσεις. Τώρα, όταν εσείς ε, μιλάτε για τη δημιουργία μιας ε, ενό ευρωπαϊκού οργανισμού, μια ευρωπαϊκή αρχή. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται η δημιουργία άλλου ενό οργανισμού. Ανταυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να διευκολύνει τον καλύτερο συντονισμό της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Επίσης πιστεύουμε ότι μία βάση δεδομένων ε, σχετικά με την παράνομη εργασία θα ήταν εφικτή. Χρειάζεται όμως πάρα πολύ καλό συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πιστεύω πως σε βάση πρέπει να δώσουμε στην, στον μη σεβασμό των συνθήκων εργασίας και όχι στις εκκυρώσεις των μεμονωμένων δραστηριοτήτων, ε, παράνομων δραστηριοτήτων στα κράτη-μέλη. Επίσης, καλωσορίσουμε την ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης, διότι πιστεύουμε ότι διευκολύνει τις διασυνοριακές επιθεωρήσεις εργασίας. Είναι μια κάρτα με, που είναι θελοντική και ε, πιστεύουμε πως θα έπρεπε να είναι εθελοντική και όχι υποχρεωτική, γιατί πιστεύουμε πως θα έπρεπε να θεωρεί ο κάθε εργαζόμενος ότι είναι προς το δικό του συμφέρον να έχει μια τέτοια κάρτα όταν εργάζεται στο εξωτερικό. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιθυμούσε η Επιτροπή να προσθέσει κάτι, όχι, ή η η έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Όλα τα σχόλια είχαν να κάνουν ε, με την ε, αποφυγή του, των εθνικού προστατευτισμού με την ε, άρση των εμποδίων. Να σας πω ότι η νομοθεσία δεν είναι καινούρια. Δεν ζητούμε κάτι καινούργιο, ζητούμε απλά να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, την καταπολέμηση της ε, παρανομίας και της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή αργορά εργασίας, ε, στην οποία όμως, ε, την οποία όμως αντιμετωπίζουμε με εθνική νοοτροπία. όταν ακούω από τις εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας ότι δεν είναι σε θέση να επεξεργαστούν τα δεδομένα που έχουν, τότε αυτό καθιστά σε εμένα τουλάχιστον προφανές ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή αρχή επιθεώρησης εργασίας. Πιστεύω ότι το πρόβλημα ε, οφείλεται στις διαφορές ε, του συστήματος επιθεώρησης εργασίας στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και χρειάζεται μια δημιουργία ευρωπαϊκής Κεντρική Αρχή Τώρα, όσον αφορά το βελγικό σύστημα που αναφέρθηκε, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε και πιστεύω πως αν διαβάσετε πολύ καλά την απόφαση θα δείτε ότι δεν ασκεί κριτική στο σύστημα λιμόζα αλλά την ε, αντιμετώπιση των αυτοαπασχολούμενων από άλλα κρατημέλη από τρίτες χώρες. Το βελγικό κράτος εισήγαγε το σύστημα αυτό διότι ήθελε να αποτρέψει την ε, καταστρατήγηση του νομικού πλαισίου όσον αφορά την αυτοαπασχόληση ή την ψευδή αυτοαπασχόληση. Δυστυχώς όμως ασκήθηκε κριτική ακριβώς σε αυτό το ε, σημείο της ε, βελγικής ε, απόφασης. Όμως είμαι σίγουρη πως θα βρούμε κάποιο κοινό παρονομαστή με του υπόλοιπου κοιόδη εισηγητέ, διότι το ζητούμενο είναι να βοηθήσουμε τους εργαζόμενου. ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία εισηγήτρια θα εξετάσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στη συνεδρίασή μας της 25ης Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε την επόμενη μέρα και την έκθεση συνολότης. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης. Φτάνουμε στο σημείο 14. Δίνω το λόγο εκ νέου στη Γιούτα Στάινλουκ να εξετάσουμε την εξουσδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν προ τη συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση Διεθνού Οργάνωση Εργασία του 1990 για την ασφάλεια κατά τη χρησιμοποίηση των χημικών προϊόντων στην εργασία. Κυρία εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Μάλιστα, α ε, την πούμε εν συντομία σε σύμβαση ήλιο, σύμβαση του ΠΟΕ. Χαιρετίζω λοιπόν την πρόταση για απόφαση του ε, Συμβουλίου να δοθεί δυνατότητα στα κρατη να κυρώσουν την ε, σύμβαση αυτή, την σύμβαση 170. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να κυρώσουν από μόνα τους ε, την, ε, την σύμβαση αυτή χωρίς την ε, σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. Και η σύμβαση αυτή ήδη μέσω του κανονισμού REACH ή του κανονισμού ταξινόμησης, επισήμανσης και ε, συσκευασίας των χημικών εφαρμόζεται. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη. Πιστεύω πως με την κύρωση της ε, συμφωνίας, ε, της σύμβασης αριθμός 170 θα ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας κατά τη χρήση χημικών προϊόντων. Και στηρίζω λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξουσιοδότηση κύρωση και ελπίζω να υπογράψουν την σύμβαση αυτή όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη. Ε, Σας ευχαριστώ. Ο κ. Καλτσίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω μερικά λόγια εκ μέρους του συναδέλφου Μπάνιον. Έχει μια ομάδα επισκεπτών, βλέπετε, και είναι από αυτή τη φάση. To add is, ε, αυτό που ήθελε είχε να συμφωνήσουμε εν γέννη με την προσέγγιση της εισηγήτριας. Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι χρηματοδότης έχουν διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά μέσα. Συγγνώμη, λέει ο μιλήτης. Sorry, it's not that report. Sorry. Ε, έκθεση. Συγγνώμη. Alors, euh, sur la 170 όσον αφορά τη χημεία. Για την 170 σύμβαση υπάρχει κάποιος το λόγο, δεν υπάρχει. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Θα τεθεί προθεσμία για τις τροπολογίες μόνο στα αγγλικά, για, μόνο για το νομοθετικό ψήφισμα, για τη σύσταση. Μπορούμε να πούμε ναι ή ου, 7 Νοεμβρίου στις 12 είναι η προθεσμία. Θα εξετάσουν τις τροπολογίες 14 Νοεμβρίου και θα ψηφίσουμε ως συνήθως στη διαδικασία. Τελειώσαμε αυτό το σημείο. Η Αντιπρόεδρος είναι Σούμπερ, έχει το λόγο για να αναφερθεί στην άλλη σύμβαση της ημερήσιας διάταξης. Την 189 κινητοποιηθήκαμε για αυτό το θέμα. Δηλαδή, εξουσιοδότηση των κατών μελών ακυρώ του συμφέροντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση Διεθνού Οργάνωση Εργασία 2011 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό. Η κυρία Σιγήτρη, κυρία Ζούμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. κύβευμα έγκυται στην προστασία των εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι περισσότερο από τους άλλους εξαιτίας της εργασίας τους και όπου κατά την εργασία είναι απομονωμένοι. Πέρα από αυτό γνωρίζουμε σήμερα ότι ότι περισσότεροι που ανήκουν σε αυτή την ευάλωτη κατηγορία είναι γυναίκες ή ε, διακινούμενοι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι αυτοί δεν γνωρίζουν καν τα δικαιώματά τους, το ότι έχουν και εκείνοι, διαθέτουν και εκείνοι δικαιώματα, όπως και όλοι οι άλλοι, και ότι βρίσκονται στο και στην ουσία βρίσκονται στο χέρι των εργοδοτών πολλές φορές αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, ακόμα και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, βίας και συμμετέχουν στα δίκτυα δουλεμπορίου και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύμβαση αυτή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, όπως είπε και η πρόεδρός μας, και ορισμένες πτυχές της σύμβασης αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ελευθερία μετακίνησης ή διακίνησης και γι' αυτό το, τα κράτη-μέλη πρέπει να κυρώσουν τη σύμβαση. Εάν λοιπόν επέλθει συμφωνία με βάση τη σύσταση που προβάλλω, τότε θα επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν χώρες από όπου προέρχονται οι μεταναστευτικές αυτές ε, ροές που έχουν κυρώσει συμφωνία όπως Μαυρίκιος, Νικαράγουα και άλλες χώρες. Και αυτό που έχει σημασία αναγνωρίζονται δικαιώματα όπως ε, συμμετοχή στις συλλογικέ διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και ούτω καθεξής, συμμετοχή στα συνδικάτα κλπ. Επίσης μιλάμε για κατόφλια τα οποία θα πρέπει να ε, τηρούν τα κράτη-μέλη και, εν πάση περιπτώσει, οι οικιακοί εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να στερούνται των δικαιωμάτων τους. Πολλές φορές ε, μένουν στο σπίτι του εργοδότη, κατοικούν εκεί και δεν ε, τηρούνται, δηλαδή δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους ως προς την ξεκούραση, το δικαίωμα σε άδεια, διακοπές και ούτω καθεξής. Επίσης η σύμβαση αναφέρεται σε πληροφορίες για τους, για κατοίκων αυτούς εργαζόμενους και Τη στιγμή που προσλαμβάνονται οι μετανάστες αυτοί θα πρέπει να, έχουν, να διαθέτουν μια γραπτή σύμβαση. Και μέσα στα πλαίσια της ελεύθερης διακίνησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα δικαιώματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να γίνει έλεγχος του δουλεμπορίου ιδιαίτερα, που αφορά ιδιαίτερα τις ε, γυναίκες και ας μην προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ε, μιλάμε για ε, δικαίωμα στην εξεκούραση, στην αποχή από την εργασία, μέσα στο 24ωρο, μιλάμε για έναν ελάχιστο μισθό και υπάρχει μια σειρά τέλος πάντων εγγυήσεων που προβλέπονται από τη σύμβαση. Στην αιτιολογική έκθεση επισύρω την ε, ε, προσοχή στα δικαιώματα των εργαζομένων και στο γεγονός ότι θα πρέπει να καλύπτονται τα δικαιώματα των κατοίκων εργαζομένων, διότι πρόκειται για μια ε, κατηγορία που είναι πιο ευάλωτη από άλλες. Η πρόταση ψηφίσματος ε, λαμβάνει υπόψη και την σύσταση του Συμβουλίου για κύρωση αυτής της ε, σύμβασης, κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη. Ζητά κάποιος το λόγο. ο κύριος Ουγγουράνο. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Να πω ότι πράγματι Πιστεύω ότι το εμπόριο ανθρώπων, το να παρασύρονται οι άνθρωποι μέσω αυτής της καταστάσεις, υποταγής, υπό το πρόσχημα οικιακής εργασίας, είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Νομίζω ότι η σύμβαση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας είναι καλή βάση. Δοθέντως αυτού, η ομάδα μου το ΕΛΚ θα υποστηρίξει πλήρως ε, την έκθεση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου. Και μετά κυρία Κοστέλο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να πω ότι εκ μέρους των σοσιαλιστών συμφωνούμε. Θέλουμε να προχωρήσει η πρόταση. Χρειάζεται να έχουμε ελάχιστη προστασία των εργαζομένων οπότε να τους προστατεύουμε αυτούς τους ανθρώπους σε εποχές οικονομικής κρίσης. Πολλές περικοπές γίνονται δύσκολη καιρή και οι οικιακοί εργαζόμενοι είναι οι πιο ευάλωτοι, από τους πιο ευάλωτους. Σωστά το λέει στην επεξηγηματική έκθεση ότι σύμφωνα με τη Eurostat 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτήν την κατηγορία έχουμε, οι περισσότερες είναι γυναίκες. Οι μισές είναι μετανάστρες, είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, μεγάλης εκμετάλλευσης, είναι επισφαλείς συνθήκες εργασίας, χαμηλές οι αμοιβές, Πολλέ πολλές ώρες εργασίας, καμιά φορά είναι θύματα σεξουαλικής βίας, εμπορίου, εκμετάλλευσης. Πρέπει να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε τις συμβάσεις τους, να υπάρχει πλήρης προστασία των δικαιωμάτων τους, των κοινωνικών και άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, νομίζω ότι πρέπει να προωθήσουμε το θέμα αυτό Πιστεύουμε ότι η αξιοπρεπή εργασία είναι το κλειδί για την εκρίζωση της ένδειας, για τη βελτίωση της ζωής ανδρών και γυναικών, για τη σταθεροποίηση της οικονομίας και να μπορούν με αξιοπρέπεια να ζουν οι άνθρωποι και ειρηνικά. Σαν πολιτική ομάδα λέμε ότι η αξιοπρεπή εργασία είναι η βάση για την αξιοπρεπή ζωή. Είμαστε θετικότατοι λοιπόν όσον αφορά την άδεια, την έγκριση που θα δοθεί στα κράτη-μέλη να κυρώσουν προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης την σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σχετικά με την εξωπρεπή εργασία του οικιακού προσωπικού. Σας ευχαριστώ, κυρία Κοστέλο. Βάσει των όσων υπόθηκαν, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι καλό να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση 189. Η εξωπρεπής εργασία ε, του οικιακού προσωπικού προστατεύεται αναφέρθηκαν καταχρήσεις, η βία κατά των ανθρώπων αυτών, η εκμετάλλευσή τους, δεν θα επαναλάβω όλα τα προβλήματα. Αξίζει να πούμε ότι και καργαζόμενοι κοινωνικά και οικονομικά, ε, είναι πολύ σημαντικοί για τις οικονομίες όλων των κρατών μελών. Για την ώρα όμως είναι επισφαλής εργασία, υποτιμάται και νομίζω ότι η έγκριση και εφαρμογή της Σύμβασης 189 τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία θα μετατρέψει επισφαλή εργασία σε αξιοπρεπή απασχόληση. Πρέπει να θεωρηθεί ότι η εφαρμογή τη Συμβάσεω 189 τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία πρέπει να είναι η βάση και όχι η οροφή. Και πρέπει να έχουμε στόχο τη βελτίωση των συνθήκων για το οικιακό προσωπικό και για τον σεβασμό των δικαιωμάτων του προσωπικού αυτού. Κυρία εισηγήτρια, όχι, ουδέν σχόλιον. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Λέει εισηγήτρια, δεν έχω τίποτα να πω λοιπόν. Άρα προχωρούμε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να θέσουμε προθεσμία για τις τροπολογίες αγγλικά και για το νομοθετικό ψήφισμα μόνο. Προθεσμία 7 Νοεμβρίου 2013, 12 το μεσημέρι. Όπως και για το προηγούμενο κείμενο που συζητήσαμε. Συζήτηση τροπολογιών. 14 Νοεμβρίου. Ελπίζουμε η ψηφοφορία στην Επιτροπή να λάβει χώρα την ίδια μέρα. Φτάσαμε στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης. Δίνω το λόγο στο Σέργιο Γκουτιέρες Πριότο να μας μιλήσει για το σχέδιο γνωμοδότησής του για την Οικονομική Ζωνετική Επιτροπή που αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ε, χρηματοπιστωτική κρίση αποτέλεσε μεγάλο μάθημα για μας και πολίτες καθώς και επιχειρήσεις ε, καταβάλουν το αντίτιμο. Θα πρέπει όμως ε, να βρούμε και συστήματα χρηματοδότησης και ρύθμισης μέσα στα πλαίσια μιας διαφάνειας για τις αποταμιεύσεις των πολιτών προς επενδύσεις που οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτός είναι και ο στόχος της πράσινης αυτής βίβλου, να δούμε πώς δηλαδή από τις δημόσιες αρχές να προβάλλονται πρότυπα για αποταμιεύσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακροχρόνια και τις σχετικές επενδύσεις δυνάμει της ε, στρατηγικής 2020 μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ε, ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε οι δημόσιες αρχές πώς μπορούν να προσανατολίσουν τις αγορές έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα μέσα όπως η κοινωνικής υφής επενδύσεις που αυτή τη στιγμή αποκλείονταν μέσω των ε, ε, μεσαζόντων από τους μεσάζοντες που υπήρχαν μέχρι τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε και να ενισχύσουμε μηχανισμούς που ήδη προϋπάρχουν για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους δεν έχουμε εισαγάγει όλες τις ιδέες που θα θέλαμε. Αυτό θα γίνει και μέσω τροπολογιών, αλλά σε γενικές ε, γραμμές ε, προβάλλουμε 4-5 ιδέες. Ε, βασιζόμαστε σε έναν μακροχρόνιο συμβιβασμό σε σχέση με την τάση που έχει διαγραφεί την ε, τελευταία δεκαετία, δηλαδή να μην υπάρχει ε, κερδοσκοπία, ε, να απαλληφθεί η κερδοσκοπία που ενισχύθηκε από την κρίση που ζούμε, να υποστηρίξουμε τις, και τις δημόσιες αποταμιεύσεις και τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις και να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων προωθώντας και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προωθήσουμε και τις μακροχρόνιες επενδύσεις για να φτάσουμε σε ένα επωνομαζόμενο δημιουργικό κεφάλαιο, χρησιμοποιώντας και του, τις φορολογικές διευκολύνσεις για την ε, καινοτομία και την ανάπτυξη καθώς και την έρευνα που χρειάζεται όλο ένα και περισσότερο η Ευρωζώνη. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα για να γίνει αυτή η χρηματοδότηση να προωθηθεί προς τις ε, ΜΜΕ διότι όταν συγκρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες ε, πλευρές, ε, με άλλα σημεία του κόσμου, βλέπουμε ότι υπολοιπόμαστε κατά πολύ. Σε άλλες χώρες αυτά τα προγράμματα, αυτές οι επενδύσεις προβάλλονται υπέρ των ε, ΜΜΕ. και βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, προβάλλουν αυτές, ε, τα, αυτά τα μέσα για την ε, χρηματοδότηση ή αυτοχρηματοδότηση. Επίσης, θα θέλαμε να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι να ενταχθούν στην ε, στρατηγική 2020 όπως στην περίπτωση της ε, κοινωνικής εστίας και της κοινωνικής κατοικίας γενικότερα μέσα στα πλαίσια των, ε, της στρατηγικής 2020. Θα πρέπει να υπάρξει η σωστή χρηματοδότηση με χρησιμοποίηση και ε, κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, όπως έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Να υπερασπιστούμε τις ε, ΜΜΕ. Γιατί το κεφάλαιο υψηλού κινδύνου πολλές φορές ε, χρησιμοποιείται για την υποστήριξη των ΜΜΕ, των ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες εχμής. Τα επισφαλή αυτά κεφάλαια λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπέρ των ΜΜΕ. Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούν ή προωθούν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Αυτά προβάλλει η πράσινη βίβλος για το μακροοικονομικό πλαίσιο χρηματοδότησης με βάση τα κριτήρια της ε, καλύτερης ε, χρησιμοποίησης ε, μέσων και μιλάμε και για collateral capital το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκεί όπου χρειάζεται. Νομίζω ότι αυτά τα μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν πρότυπο χρηματοδότησης και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πώς χρησιμοποιούνται ε, τα ε, χρήματα των συνταξιοδοτικών ε, ταμείων. Να, υπάρχει καλύτερη, να υπάρχουν καλύτεροι έλεγχοι από αυτούς που υπήρχαν μέχρι τώρα. Δηλαδή να αντιλήσουμε τα σωστά διδάγματα από την παρούσα κρίση για να προωθήσουμε πραγματικά μια κοινωνία ευημερίας, έτσι ώστε οι αποταμιεύσεις των πολιτών να χρησιμοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Α, αυτές είναι οι βασικές ιδέες της ε, έκθεσης αυτής. Ε, Κασίμ, ευχαριστώ. Ε, αυτή είναι η παρέμβαση που ήθελα να κάνω. Βιάστηκα όμως πιο πριν. Ο συνάδελφός μου που απουσιάζει, που έχει την ομάδα των επισκεπτών, έχει προετοιμάσει μια παρέμβαση την οποία ήθελα να μοιραστώ μαζί σα Σε γενικέ γραμμέ, σύμφωνοι με την προσέγγιση του εισηγητή για τη γνωμοδότηση αυτή, για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Είναι δύο διαφορετικοί ε, στόχοι που θα με διαφορετικά μέσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι δύο ε, αυτές οι επιτυχίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στι ίδιε περιπτώσει. Είναι ε, φανερό ότι στο μακροπρόθεσμο σκέλος πρέπει να συμπεριληφθούν ε, και άλλα πράγματα πέραν των οικονομικών επιτυχών. Μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση μπορεί να δώσει περισσότερη σταθερότητα, το οποίο θα είναι ωφέλιμο για όλους τους ενδιαφερόμενους. Επίσης, ε, συμφωνεί με την άποψη του εισηγητή για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ένα τεράστιο δυναμικό για νέες θέσεις απασχόλησης και οικονομική ανάπτυξη. Και ο ε, συνάδελφος συμφωνεί ότι τα πιθανά κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη της ανάπτυξης και πρόσβασης σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση θα καταφέρουν να ε, μειώσουν την εξάρτηση σε βράχη πρόθεσμα ε, υποστηρικτικά μέσα και να οδηγήσουν σε πιο υπεύθυνη χρηματοδότηση στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος που ζητά να παρέμβει. Δεν βλέπω. Κύριε Γκουτιέρες, θέλετε να δευτερολογήσετε. Όχι, εν αυτή η περιπτώση. Τέλεια. Αρκεί να πούμε ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογίων στα αγγλικά 11 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και τους συμβιβασμούς ε, στην συνεδρία 25-26 Νοεμβρίου. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προσχώρησης 17 Δεκεμβρίου. Εξυπακούεται η Οικονομική Ομοσπονδιακή Επιτροπή που να ψηφίσει στις 20 Ιανουαρίου. Όλα αυτά για να πάμε στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο, στη δεύτερη. Φτάσαμε στο σημείο 17. Δίνω το λόγο στον Μάρτιν Κάστλερ. Σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών. Θέμα το δίκτυο Solvit. Κύριε Ισηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχετε όλοι λάβει την πρότασή μου και πρέπει να πω ότι η συνεργασία που είχαμε όλους ήταν πάρα πολύ καλή όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος όλων μας είναι μια εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και πιστεύω ότι ε, σε αυτή την έκθεση ε, αναφέρονται κάποια πολύ σωστά σημεία. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι χρειάζεται μια ε, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Solvit, δηλαδή είναι μια διαρθρωτική σε φύση αλλαγή. το Solvit ε, επεμβαίνει και σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής ε, του ευρωπαϊκού δικαίου από τα κράτη-μέλη. Έπειτα δεύτερο τομέα, η συμπερίληψη των ε, συντάξεων. Σήμερα ακούσαμε πάρα πολλά για τις συντάξεις και πιστεύω πως και, και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα μπορούσε να επιληθεί με το πρόγραμμα Solvit. Ε, για παράδειγμα, ένα πρόβλημα είναι η ε, φορητότητα των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το οποίο συζητήσαμε πριν από λίγη ώρα. Το Solvit λοιπόν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό έτσι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ένα τρίτο σημείο είναι μια ιδέα που ε, υπέβαλα εγώ ίδιος προσωπικά και ευχαριστώ πολύ και, και για την στήριξη των συναδέλφων είναι η ιδέα του Solvit Regio, του περιφερειακού Solvit κέντρων δηλαδή που θα αναπτύσσονται σταδιακά έτσι ώστε να δώσουν στις ευρωπαϊκές περιφέρειες την ευκαιρία να ε, δημιουργήσουν αναγνωρισμένα περιφερειακά κέντρα που θα καλύπτουν τις ε, διοικητικές τους ε, ανάγκες και θα ευαισθητοποιήσουν. Πιστεύω πως έχουμε υποδομές στα κράτη-μέλη και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις υποδομές έτσι ώστε να ε, βοηθήσουμε αυτές τις ε, αποκεντρωμένες ε, μονάδες, είτε αυτές βρίσκονται σε κάποιο γερμανικό κρατήδιο, είτε σε κάποια περιφέρεια άλλου ευρωπαϊκού κράτους. Πιστεύω πως σε όλες οι γενικές γραμμές συμφωνούμε ότι το Solvit χρειάζεται να έρθει πιο κοντά στους ανθρώπους της περιφέρειας και πιστεύω πως με τον με την πρόταση αυτή με, ε, και αν έχω τη στήριξή σας ε, στην πρωτοβουλία θα μπορούμε να το καταφέρουμε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για, τις, ε, για τη συνεργασία. Θα χαρώ πολύ να λάβω τις προτάσεις σας και είμαι αισιόδοξο ότι θα καταφέρουμε να έχουμε ένα τελικό έγγραφο χωρίς προβλήματα και όλοι μαζί με τους σκιώδους εισηγητές θα μπορέσουμε να έχουμε μια πάρα πολύ συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σέρκας. Ε, εξ του κύριου, του κύριου Μπαλτακίνο που δεν ε, μπορεί να είναι εδώ, έχω εδώ μία σημείωση. Eh? Το άλλο μικρόφωνο δεν ήταν δικό μου. θα ήθελα να πω είναι ότι ο κύριος ε, ε, Μπαλτακίνο δεν είναι ε, πολύ ικανοποιημένο ως προς την προσέγγισή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι για μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για περιφερειοποίηση, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει σε θελούσια βάση, μέσα στα πλαίσια της ε, επικουρικότητας. Και με βάση τις σημειώσεις που έχω εδώ, θα ήθελα να πω ότι το, μέσον, το μέλλον συγγνώμη, βρίσκεται online, γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε το Solve It online, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πρόβλημα προσβασιμότητας στο διαδίκτυο. Θα συνεργαστούμε μαζί σας ε, για να προωθήσουμε θέματα που αφορούν το, το συμφέρον των πολιτών και της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Κιόδους της Μέρι Χάρκιν για τους φιλελεύθερους θα ήθελα ε, να μιλήσω και να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το πολύ καλό έγγραφο. θεωρώ την ε, λύση του Solvit Regio της ε, περιφερειοποίησης, δηλαδή του δικτύου Solvit, πάρα πολύ καλή. Επίσης ε, μπορούμε να στηρίξουμε και την πρόταση για συμπερίληψη όσο το δυνατόν περισσότερων ομάδων και περισσότερων υπηρεσιών για τους πολίτες. Επίσης, η Mary Harkin θεωρεί το προσχέδιο ήδη πάρα πολύ καλό. θα υποβάλει ωστόσο έναν μικρό αριθμό τροπολογιών έτσι ώστε να τελειοποιηθεί το έγγραφο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, επιστρέφω και δίνω τον, ρόλο στον τον λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη και για τα θετικά σας λόγια. Πιστεύω πώς θα καταφέρουμε ε, το έργο που έχουμε αναλάβει. Είναι σχεδόν τέλειο. Εγώ πιστεύω πως είναι ήδη τέλειο, κυρία Πρόεδρε, αλλά ελπίζω να έχουμε έτσι μια βαβαρική αλληλεγγύη μεταξύ μας. Πραγματικά πιστεύω πως έχετε δίκιο, πρέπει να συμπεριληφθεί η διαδικτυακή διάσταση και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να την συμπεριλάβουμε. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ για την επικείμενη καλή συνεργασία. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Θα ήθελα τώρα να, ζητή, να ρωτήσω κάποιον από την ΓΔ Μάρκα, την Ανούσκα Γιάντσεν, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συντομότατα, καταρχάς να αναφερθώ σε κάποιες προκλήσεις που βλέπουμε τα επόμενα χρόνια για το Solvit και κάποιες εξηγήσεις να δώσω για τα θυγέντα θέματα. Αυτά που αναφέρθηκαν πριν από δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα, βασικές προκλήσεις είναι να έχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών παρά τους περιορισμούς των κονδυλίων και τους περιορισμούς ανθρώπινους πόρους αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να είμαστε αποδοτικότεροι στο μέτρο του δυνατού. Και χρειαζόμαστε βέβαια επαρκείς ανθρωπίνους πόρους να συνεχιστούν οι πιέσεις και ευχαριστούμε πάντα για την υποστήριξή σας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τις πιέσεις που ασκείτε προς τα κάτι μέλη γι' αυτό. Μετά πρέπει να θυγαμιστούμε με άλλα μέσα και διαδικασίες. Έτσι μπορούμε να είμαστε αποδοτικότεροι και να εξασφαλίσουμε ότι ακόμα και εκείνοι που δεν μπορούν να βοηθηθούν από το Solvit μπορούν να απευθύνονται προς τα εκεί που μπορούν να έχουν βοήθεια. Διότι δηλαδή, το Solvit δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Το Solvit αφορά παραβίαση δικαίου κοινοτικού από δημόσιες αρχές σε ένα κράτος μέλος. Είναι σημαντικό κριτήριο νομίζω να είναι υπόψη για το τι μπορεί να κάνει το Solvit. Είναι η βάση του Solvit. Δηλαδή τα κράτη-μέλη υποχρεώνονται να εφαρμόσουν σωστά το ευρωπαϊκό δίκαιο και γι' αυτό τα κέντρα Solvit είναι στις κεντρικές κυβερνήσεις και είναι ένα τμήμα της κεντρικής κυβέρνησης. Τρίτον, εξίσου σημαντικό, το κέντρο Solvit πρέπει να χρησιμοποιεί την υφιστάμενη γνώση, εκεί, αν υπάρχει και σε άλλο κράτος μέλος, να χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις. Καλούμε λοιπόν τα κέντρα Solvit των κρατών μελών να έχουν αγαστή συνεργασία με τα εθνικά μέλη της Διοικητικής Επιτροπής για το συντονισμό σε θέματα κοινωνικής ε, πρόνοιας. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι, οι περισσότερες υποθέσεις τα αφορούν την κοινωνική ασφάλιση και συναφείς υποθέσεις και είναι ένα από τα αιτήματα που είχατε κάνει στο σχέδιο γνωμοδότησής σας όσον αφορά τις συντάξεις και ξανά εκεί πέρα, από τη στιγμή που υπάρχει παραβίαση ε, κοινοτικού δικαίου, μπορεί να βοηθήσει το Solvit, αλλά χρειάζεται παραβίαση του κοινοτικού δικαίου για να γίνει κάτι τέτοιο. Άλλη μεγάλη πρόκληση. Πρέπει εκείνοι που χρειάζονται το Solvit να το βρίσκουν. Και δεν σημαίνει ότι θέλουμε 510 εκατομμύρια άνθρωποι να ξέρουν τι είναι το Solvit. Θέλουμε ο καθένας από τα 510 εκατομμύρια τη στιγμή που θα αντιμετωπίζει πρόβλημα να απευθύνεται προς το Solvit και εκείνη τη στιγμή να το βρίσκουν το Solvit όταν θέλουν. Και ένας από τους τρόπους να το πετύχουμε αυτό είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος έχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες, τα δικαιώματα που προκύπτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έρχεται και στο πύλη Europe που λέγεται που αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν την Ευρώπη. Είναι εύκολε πληροφορίε, εύληπτες, ρεαλιστικές και ο κόσμος άμα ξέρει τα δικαιώματά του ξέρει και πότε παραβιάζονται αυτά και μπορεί να προσφύγει στο Solvit. Λοιπόν, βασιζόμαστε στις ενδιάμεσες τοσελίδες, στις ενδιάμεσους φορείς, να μπορούν να επισημάνουν στον κόσμο ότι μπορούν να απευθυνθούν στο Solvit για βοήθεια. Και τελευταίο μου σχόλιο, που αφορά την κατάσταση σε περιφερειακά, στα περιφερειακά γραφεία του Solvit, ενθαρρύνουμε τα μάλα τα κέντρα Solvit να γνωστοποιούν τη θέση τους στις τοπικές αρχές και περιφερειακές αρχές, ούτω ώστε αυτοί οι φορείς να δρουν ως ενδιάμεση. Όταν χτυπάει την πόρτα ένας πολίτης περιφερειακής αρχής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, με ένα πρόβλημα που μπορεί να επιληθεί από το Solvit, να γνωρίζουν τι είναι το Solvit και να κατευθύνουν αυτούς τους ανθρώπους προς το Solvit. Αυτά είχα να πω, αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, thank you. Καλώ, σας ευχαριστώ εγώ. Προθεσμία 12 Νοεμβρίου για υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Επασχόλησης στις 17 Δεκεμβρίου. Άρα χριστουγεννιάτικο δωράκι. Αυτά. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, ε, βέβαια, το 18. Υπάρχουν εργαλεία για την παρακολούθηση αποτελεσματικότητα των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για του εργαζομένου μεγαλύτερη ηλικία. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Ντανούτα Γιασλιοβεύσκα. Είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτή όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης. Δίνω το λόγο λοιπόν στην Ντανούτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα θέλω να πω ότι ήδη του χρόνου θα δούμε μια μείωση του αριθμού των εργαζομένων ηλικιωμένων. Η γυράσκουσα μάλλον κοινωνία θα γίνει πραγματικότητα. Και τα κίνητρα για πρόρηση ταξιοδότηση λόγω της οικονομικής κρίσεως και της λες απαιτήσει για δεξιότητες των εργαζομένων είναι πράγματα που θα επηρεάσουν αρνητικά τον αριθμό των επαγγελματικά δραστηρίων ε, πολιτών. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο 50% των ατόμων 55 μέχρι 65 εργάζονται. Άρα η δική μας κατάσταση επιδεινώνεται από ότι σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία. Εκεί πάνω από 60% της ηλικιακής αυτής ομάδας είναι ενεργή. Υπάρχει τεράστια επιρροή, επίδραση της οικονομικής κατάστασης κράτη-μέλη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν πολύτιμη εμπειρία στον τομέα εργασίας και έχουν και την προθυμία να εργαστούν περισσότερο. Πρέπει να δημιουργήσουμε τι προποθέσει να του ενθαρρύνουμε να παραμείνουν ενεργοί. Το να κάνουμε του ηλικιωμένου πιο δραστήριου ήταν μια από τι βασικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η στρατηγική τη Λισαβόνα αναφέρεται στην ανάγκη παράταση των δραστηριοτήτων με σχέση, με σχέση εργασιακή και οι στόχοι του 2020 περιλαμβάνουν φιλόδοξο στόχο του 75% απασχόλησης των ανθρώπων αυτών της ηλικίας αυτής μέχρι 64 ετών δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς οι πιο ηλικιωμένοι να συμμετάσχουν. Ήδη από το 1957 βασικό εργαλείο που είχαμε στη διάθεσή μας, η συγκριματοδότηση και η δράση που έχουν στόχο την αγορά εργασίας και ε, εργασιακές δραστηριότητες που συμπραβάνουν τους ηλικιωμένους είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Το 2007 με 2013 75 δισεκατομμύρια ευρώ δόθηκαν στο Ταμείο, αυτό σημαίνει 80% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν 117 επιχειρησιακά προγράμματα, 63 από αυτά τα λειτουργικά προγράμματα είχαν σαν στόχο άμεσο ή έμεσο ε, τους πιο ηλικιωμένους εργαζομένους. Δυστυχώς, σαν, όπως δείχνει η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου του 2012, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να πούν πόσοι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι ε, στηρίχθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία, πόσοι πόροι διατέθησαν και σε ποιο βαθμό οι δράσεις ήταν αποτελεσματικές και επέτρεψαν την αύξηση των προσόντων ή την εξέβρεση νέων θέσεων απασχόλησης από πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους. Μόνο στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας και του Γιβραλτάρ οι πληροφορίες όσον αφορά ε, τους πιο ηλικιωμένους ήταν διαθέσιμα. Η έλλειψη στοιχείων οφείλεται στη μη εφαρμογή των σωστών μέτρων ελέγχου και την επιλογή των ποιοτικών α, δικτών που είναι κατάλληλοι. Είναι θαρρυντικό διότι στο μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ο κανονισμός για τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία συμπεριλαμβάνει διόρθωση των εργαλείων αξιολόγησης για αποδοτικότητα των προγραμμάτων και εισάγει ένα, μια ομάδα δικτών που έχουν σαν στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Στη γνωμοδότηση που παρουσίασε ενθάρρυνα επίσης τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τέτοιους δείκτες οι οποίοι θα δείκτουν επακριβώς πόσοι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι απέκτησαν νέες, νέα προσόντα, βελτίωσαν την κατάστασή τους στην αγορά εργασίας ή βρήκαν νέες δουλειές χάρη στα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Ταμεία. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις αποτελεσματικότερες δράσεις στο μέλλον. Στην έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επίσης αναφέρεται στην έλλειψη ενιαίου ε, φάσματος ηλικίας, ορισμού του ηλικιωμένου εργαζομένου. Τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά όρια, 45 συν, 50 συν ή 55 συν. Αυτό πορεύει από διαφορές κοινωνικο-οικονομικές. Για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τις δραστηριότητε που πραγματικά ανταποκρίνουν τις ανάγκες πιο, των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, Χρειάζεται ανάλυση αναγκών σε κάθε κάτω μέλο Για τις ίδιε ηλικιακέ ε, ηλικιακό, φάσμα όπως τα προγράμματα και οι δράσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε δύο ηλικιακές ομάδες και να προσαρμόζονται οι δράσεις στις ανάγκες των νέων, 45-55, κατάρτιση, απόκτηση προσόντων αυτοαπασχόληση και τις μεγαλύτερες ομάδες, 55 συν, ευέλικτη απασχόληση Φερρυπίν. Στις τροπολογίες που κατέθεσα έχω κάποιες τέτοιες ιδέες που αναφέρω, αλλά ε, υπήρχαν και κάποια όρια που μου είχαν τεθεί. Ελπίζω να ακούσω τα σχόλιά σας και ελπίζω ότι θα έχουμε καρποφόρα συνεργασία με τους κοιόδης ηγητές. Ελπίζω αυτή η γνωμοδότηση να αποτελέσει μια καλή εφετηρία για τις συζητήσεις μας. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Άλλος θέλει να παρέμβει. Otherwise... να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμμανουέλ Γκουενόη έχει το λόγο η κυρία Εμμανουέλα. Νομίζω ότι η Επιτροπή θα ήθελα να τονίσει, όπως είπατε και εσείς, ότι πολλές από τις συστάσεις έχουν ληφθεί υπόψη για την νέα περίοδο προγραμματισμού στο νομοθετικό πλαίσιο που αυτή τη στιγμή συζητάμε. Μιλάμε λοιπόν για μια συγκεκριμένη ε, στοχοθέτηση έτσι ώστε να έχουμε και μια καλύτερη αποτίμηση των επιδόσεων γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ε, πώς μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν ορισμένες πτυχές που μας απασχολούν ιδιαίτερα και που θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή ως προς την συνολική διαχείριση και θα ήθελα να πω εδώ ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει ε, πολύ καλύτερη αποτίμηση της όλης διαδικασίας. Ευχαριστώ. 13 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 21 Ιανουαρίου του χρόνου. Είναι 7 ε, και 5. Θα πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίαση. Έχουμε και το σημείο υπαριθμών 21 εδώ βλέπετε την έκθεση της αντιπροσωπείας στο Λονδίνο, στο φάκελό σας, για να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης, ε, τους αποσπασμένους, τα δικαιώματα και την εφαρμογή της ε, πραγματικής ε, προστασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα στην, ε, στο φάκελό σας βλέπετε τον, την πλήρη έκθεση. Αυτό είναι και το τελευταίο θέμα. The next... Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 14 Νοεμβρίου από τις 9 στις 12.30 στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.